Καλημέρα, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε, παρόλο που δεν είναι ακόμα η προσέλευση. Λυπάμαι, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Τζούβα, ο Σκιώδης, νομίζω ότι είχε αλλάξει τα σχέδιά του, όταν ανακοίνωσε τις πρώτες αλλαγές χθες. Ελπίζω να έχουμε κάποιον από το ΕΛΚ. Την κυρία Ιγκουάν να καλωσορίσουμε που θα μας παρουσιάσει κάποιες από τις σκέψεις της για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, την οποία η Επιτροπή και οι συντονιστές ανέθεσαν και προγραμμάτισαν και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο τομέα αυτό. Έχετε ήδη εκθέσει τις ιδέε σα για τη στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών και έχουμε και κάποιου σκιώτες μαζί μα. Ο κύριο Σμιτ δεν είναι εδώ. Η κυρία Πραβάνοβα θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Σμιτ. Τον κύριο Τεντεφολίδη να καλωσορίσω. Και εγώ θα είμαι σκιώτης από πλευρά τη ομάδα μου. Και όποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν. Ο κυρία Τουρμπλουμ είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και έχει παρακολουθήσει στενά το θέμα αυτό και με τον κύριο Μικόλα. Θα σας δώσω λοιπόν και εσάς το λόγο. Χαιρόμαστε επίσης που έχουμε εκπροσώπους της Πολωνικής Προεδρίας μαζί μας. Πολύ θετικό και αυτό. Επίσης να καλωσορίσω ιδιαίτερος τον κύριο Ανδρέα ε, Σαλτέλη από το JRC. Ομόλογός μου ε, σε άλλες δραστηριότητες της ΣΤΟΑ η οποία ε, προωθεί την ιδέα συνεργασίας βουλευτών με επιστήμονες στα πλαίσια κοινή Επιτροπής Έρευνας. Πρόκειται λοιπόν για το JRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι στατιστικό λόγος λοιπόν ο συνάδελφος. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Κυρία Ιρουγκάν Πέρες, να ακούσουμε καταρχάς τις ιδέες σας. Buenos días, buenos días a todos y muchas gracias. Καλημέρα σε όλους. Και ευχαριστώ που ξυπνήσατε τόσο νωρίς να σας δώσω κάποιες ιδέες για το θέμα της ενίσχυσης των ευάλωτων καταναλωτών. Όπως γνωρίζουμε, οι αξίες της προστασίας των καταναλωτών και η ευημερία τους αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη επίσης των στόχων της Ευρώπης 2020. Όμως μέσα στο, σε όλους τους καταναλωτές υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών, αυτούς που αποκαλούμε καταναλωτές σε κατάσταση ευάλωτη και που χρειάζονται μια ειδική στρατηγική από πλευρά των αρχών. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η έκθεση δεν προσπαθεί να δώσει κάποιον ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ιδέα αυτή του ευάλωτου καταναλωτή. Δεν θέλουμε ωστόσο να είναι εξαιρετικά όρεστη, εξαιρετικά συγκεκριμένη, χωρί την απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται στις ε, ειδικέ συνθήκες που μπορεί να πλήξουν ένα τέτοιον καταναλωτή. Δηλαδή μπορεί όλοι μας να βρεθούμε σε αυτή την ευάλωτη θέση ε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, διότι αυτή η κατάσταση καθορίζεται από ενδογενείς ή από εξωγενείς παράγοντες. Ενδογενείς μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες αιτίε που είναι ενδογενείς της κατάστασής του, της σωματικής ή της ψυχικής, είτε πρόκειται για παιδιά, για εφήβους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ηλικιωμένους ανθρώπους και εξωγενείς παράγοντες είναι αυτοί που οδηγούν έναν καταναλωτή σε ευαίσθητη θέση, έλλειψη γνώσεων, έλλειψη γλωσσικών γνώσεων ή το γεγονός ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες τις οποίες δεν γνωρίζει απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε πως η νομοθεσία η ευρωπαϊκή για πρώτη φορά μιλά για το καταναλωτή στην οδηγία του 2005 σε σχέση με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων σε σχέση τους με τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά θεσπίζοντας μια ε, έννοια προσαρμοσμένη σε αυτές τις πρακτικές με επίκεντρο την ε, αθέμητη επιρροή που μπορεί κανείς να ασκήσει σε έναν καταναλωτή. Ωστόσο, αυτή η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές προστατεύει μόνο τα συμφέροντα των καταναλωτών και όχι, δεν καλύπτει άλλους τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια ή η ηθική κυριότητα. Η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που είναι το πιο πρόσφατο μέσο που είναι αφιερωμένο στην προστασία του καταναλωτή, κατά τη γνώμη μου αφορά ε, συγκεκριμένες ε, απόψεις ε, των Νοέμβριο του 2005 η Κομισιόν εξέδωσε ανακοίνωση με στόχο την ενίσχυση του καταναλωτή ώστε να μπορέσει να εδρεώσει τα δικαιώματα του καταναλωτή και να ενισχύσει τα δικαιώματα προσφυγής αλλά και τον έλεγχο του σεβασμού των δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. Χαιρετίζω τη φιλόδοξη αυτή προσέγγιση της Κομισιόν και ο κανονισμός αυτός διευκρινίζει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων καταναλωτών, να λάβουμε υπόψη την κατάστασή τους και όλος ιδιαίτερος την κατάσταση των ηλικιωμένων ανθρώπων καθώς και την κοινωνική τους ένταξη, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι αυτόνομοι φορείς στην αγορά και το δίδυμο ευάλωτοι καταναλωτέ και τρίτη ηλικία τονίζεται όλο ιδιαίτερο, πράγμα το οποίο μπορεί να καταλήξει σε λάθη. Κατά τρίτο λόγο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κομισιόν θέλει να υιοθετήσει μέτρα σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή. Πρόκειται όμως για μια προσέγγιση που βασίζεται στο γεγονός ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες εξουσίες στον ίδιο τον καταναλωτή και άρα πρέπει αυτός να είναι πιο αυτόνομος, πιο ανεξάρτητος και αυτό γίνεται μόνο μέσω της γνώσης των δικαιωμάτων που έχει ο ίδιος ο καταναλωτής. Γι' αυτό και θέλει η Κομισιόν να αυξήσει την ενημέρωση, να ενισχύσει την ενημέρωση προς τον καταναλωτή, ώστε να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του, αλλά δυστυχώς η προσέγγιση αυτή δεν αρκεί στο πλαίσιο των ευάλωτων καταναλωτών. Όντως, ο ευάλωτος χαρακτήρας πολλών καταναλωτών προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ε, είναι ακόμα, δεν, είναι, δεν έχουν απόλυτα σωστή κρίση. Δηλαδή τα παιδιά οι ηλικιωμένοι δεν καταλαβαίνουν απόλυτα καλά τις πληροφορίες που, του δίδονται, που τους δίνονται. Ε, όπως επίσης και τα αποκλεισμένα άτομα, κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, δεν κατανοούν τις πληροφορίες που τους δίνουν πάντοτε, ούτε γνωρίζουν τα δικαιώματα προσφυγής που έχουν έχουν δεν γνωρίζουν τις ισχύουσες νομοθεσίες, ιδιαίτερα σε θέματα διασυνοριακού εμπορίου και online εμπορίου. Κάθε καταναλωτή σε κάποια στιγμή της ζωής του μπορεί να, γίνει, να βρεθεί σε ευάλωτη θέση και η αυτονόμηση δεν αρκεί για να προστατευτούν τα δικαιώματά του και γι' αυτό κυρίες και κύριοι βουλευτές οφείλουμε να απαιτήσουμε από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα που να εγγυώνται κατάλληλη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών πέρα από τη συγκεκριμένη ενημέρωση για τα θέματα ή το επίπεδο, όπου το επίπεδο μάλλον ε, της βοήθειας πρέπει να είναι πιο σημαντικό, δηλαδή πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη, ε, διατροφή, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και διάφορα άλλοι τομείς. Θα πρέπει να φτιάξουμε τέτοιο είδους νομοθεσία που να λαμβάνει υπόψη τα άτομα που βρίσκονται σε πιο εύθραυστη κατάσταση και να του ενημερώνουμε, αλλά επίσης να ενημερώνουμε τους προμηθευτέ σε αυτά τα προγράμματα, ώστε να φτάσουμε σε μια συμβατική ε, ισορροπία η οποία να είναι λιγότερο αδιαφανής. Να τονίσω επίσης ότι αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε δύο διαφορετικά επίπεδα προστασίας, ε, δηλαδή παρά τις νομοθετικές ε, προσπάθειες ε, που καταβάλαμε τα τελευταία χρόνια για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, η κατάσταση των ε, ε, ευάλωτων καταναλωτών πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και περισσότερο από ό,τι έχει προσεχθεί μέχρι στιγμή. Οι περισσότεροι καταναλωτέ, το έλεγα και προηγουμένω, κάποια φάση τη ζωή του μπορεί να βρεθούν σε ευάλωτη θέση και γι' αυτό και πρέπει να προβλεφθούν προστατευτικέ νομοθεσίε, ιδιαίτερα για αυτού του είδου του καταναλωτέ. Η προστασία αυτή θα τους βοηθήσει να ενταχθούν καλύτερα και κοινωνικά και έτσι να προδεύσουμε προς μια εσωτερική αγορά πιο δυναμική και πιο ανταγωνιστική και προς μια κοινωνία πιο δίκαιη. Ελπίζω πως η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τους ευάλωτους λοιπόν καταναλωτές στις προτεραιότητες της ατζέντα για την προστασία του καταναλωτή. Τώρα, έχουμε το χρονοδιάγραμμα ως εξής. Υποβολή της έκθεσης τον Ιανουάριο του 2011, 24-25 Ιανουαρίου, προθεσμία υποβολή τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου 2012 και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 28 Φεβρουαρίου 2012 και έγκριση στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Μάρτιο κανονικά. Βασίζομαι λοιπόν στη δική σας συνεργασία Αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα βασίζομαι στους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους ήδη κάναμε μια σύντομη εισαγωγική συνεδρίαση ώστε να καταλήξουμε σε μια συμπαγή έκθεση που να εγγυάται την προστασία των πιο ευάλωτων καταναλωτών και θα τους επιτρέψει έτσι να συμμετέχουν στην ενιαία αγορά στις καλύτερες δυνατές συνθήκες σεβόμενοι την ηρεμία τους και αυξάνοντας την ικανοποίησή τους διότι στόχος της νομοθεσίας είναι να προστατευτούν οι πιο δύναμη σε σχέση με τους πιο δυνατούς. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ που ξεκινήσατε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία να προσθέσω στα όσα λέγατε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ότι οι συντονιστές επίσης έχουν κάνει κάποιες ενημερωτικές σημειώσεις για τις πολιτικές στα διάφορα κράτη-μέλη που θα φτάσουν γύρω στα μέσα Ιανουαρίου εγκαίρως για να συζητηθούν στο πλαίσιο της εκθεσής σας. Φυσικά θα σας τις δώσουμε μόλις θα υπάρχουν, μόλις θα τις έχουμε και πιστεύω πως είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση για να τροφοδοτήσει τη στρατηγική για την πολιτική για τον κατανολωτή. Ε, ο κύριος Τρενταφυλλίδης που θα μιλήσει αργότερα ήδη το έχει θίξει στην ε, δική του έκθεση. Είναι πολύ λοιπόν ε, σωστός ο συγχρονισμός στο να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τον καταναλωτή. Ο κύριος Βάμπ νομίζω θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Φιλίπ Ζουμπέ. Μετά έχουμε την κυρία Παβάνοβα και μετά θα κάνω μια μικρή συμβολή από τη δική μου ομάδα και μετά ο κύριος Τριανταφυλλίδης και η κυρία Χέτ επίσης. Ο κύριος Βάμπ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ συνάδελφε Περές για την εξαιρετική παρουσίαση των σκέψεών σας. Ξέρουμε ότι από την ομάδα σας ε, το θέμα αυτό ε, έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ και καιρό. Και πρωτού περάσω σε θέματα περιεχομένου, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Συμπάνο, ο οποίο για διάφορους ε, λόγους δεν μπορεί να παραστεί εδώ πέρα σήμερα. Θεωρούμε ότι η έννοια του καταναλωτή, του ευάλωτου, εκ πρώτης όψεως ασφαλώς και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά, σε τελική ανάλυση, η δυσκολία έγινε στο εξής ότι ο καταναλωτή που χρειάζεται προστασία θα πρέπει να διαχωριστεί με σωστό τρόπο από τον κανονικό καταναλωτή σε κάποιο τομεί. Εδώ και ο μα μας ε, θεωρεί ότι υπάρχουν πολλέ δυσκολίε που ανακύπτουν. Ε, επί της αρχής θεωρούμε ως ΕΛΚ ότι ο καταναλωτής και η καταναλωτρία δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε σε ό,τι αφορά την ίδια ευθύνη που έχει, τη δική του ευθύνη. Όταν όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει ο καταναλωτής, γιατί δεν του δίδονται για παράδειγμα πληροφορίες, γιατί υπάρχει έλλειψη διαφάνειας για παράδειγμα ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος τους. Στην περίπτωση αυτή ασφαλώς και είμαστε διατεθειμένοι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και στην έκθεση υπάρχουν σημεία όπου όντως ε, αναφέρεται ε, η ανάγκη επιπλέον προστασίας κάποιων καταναλωτών. Εκεί λοιπόν είμαστε δεδεθειμένοι να ζητήσουμε περαιτέρω βήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κλασικό ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή ορίζεται από την ηλικία, την οριμότητα, που παίζουν σημαντικό ρόλο. Θεωρώ όμως ότι ο ορισμός αυτός είναι κάπως περιορισμένος, γιατί τα προβλήματα αυτά μπορούν να ανακύψουν σε όλες τις ηλικίε ουσιαστικά, μπορούν να ανακύψουν σε όλους τους καταναλωτές. Άρα δεν ε, βλέπουμε πού ακριβώς είναι ε, η συγκεκριμένος λόγος προστασίας των καταναλωτών. Θα συνεχίσουμε ωστόσο τις επικοδομητικές ε, συζητήσεις. Θα παρουσιάσουμε και τη θέση μας σε κάθε θέμα και για το χρονοδιάγραμμα, κυρία Περές. Συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό λοιπόν προσδοκούμε μια καλή συνεργασία για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω τη θέση του κυρίου Όλη Σμιτ, ο οποίος είναι ο σκιώδης μας. Καταρχάς, θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες του προς την θηγητρία και θα διαβάσω την ε, άποψή του. Η έννοια του ευάλωτου καταναλωτή εμφανίζεται επανειλημμένα και όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν κατηγορίες καταναλωτή οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Ένα βασικό θέμα, ωστόσο, είναι ποιος θα συμπεριληφθεί στην κατηγορία αυτή. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή με διαφανή και σαφή κριτήρια, γιατί το ευάλωτο του καταναλωτή έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Την δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών και την ικανότητα λήψης υπεύθυνων αποφάσεων βάσει των πληροφοριών αυτών. Σε περίπτωση ατόμων με κάποια αναπηρία και σε αναλφάβητους υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Ξέρουμε επίσης ότι τα παιδιά δεν μπορούν να θεωρηθεί ότι λαμβάνουν υπεύθυνε αποφάσεις. Δεν θα πρέπει όμως ορισμός του ευάλωτου καταναλωτή να ε, καταλήξει υπερβολικά ευρύς. Αυτά ευχαριστώ και θα ήθελα εξ ονόματός μου να πω ότι η χρήση της ε, λέξης ε, ευάλωτου μπορεί να, μπορεί να συνεπάγεται κάποιες δυσκολίες σε κάποιες γλώσσες, γιατί υπάρχει και διαφορετική έννοια, αν θέλετε. Μιλώντας για παιδιά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κυρίως τα παιδιά αποτελούν ομάδα στόχο σε ό,τι αφορά προσπάθειες επιρροής, σε ό,τι αφορά ε, μη υγιεινό τρόπο ε, ζωής, ε, κατανάλωσης προϊόντων μη υγιεινών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να μιλήσω κι εγώ ως και θα ήθελα να επαναλάβω ότι ανυπομονώ να συνεργαστώ με το θέμα, στο θέμα αυτό με την κυρία Πέρες. Νομίζω ότι δικαίως ε, υπέδειξε ότι κατά πάσα πιθανότητα όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας να είμαστε ευάλωτοι καταναλωτές. Και φυσικά, όντας και το θέμα του πληθυσμού που γυράσκει, υπάρχουν και άλλες πολιτικές σε ό,τι αφορά τη γύρανση του πληθυσμού. Άρα να έχουμε υπόψη ότι είναι διαφορετικές οι διαφορετικοί οι όροι και διαφορετικές οι συνθήκες συμμετοχής στην, κοινωνία. Είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, θεωρώ. Να είμαστε προσεκτικοί, γιατί γνωρίζουμε ήδη, όπως είπε η κυρία Περές, ότι στη δουλειά μας ως Επιτροπή, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ε, υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους όρους των συμβάσεων, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων και εξετήσαμε θέματα όπως ο χάρτης για την ενέργεια, θέματα μεταφορών και το καθεξής. Άρα θεωρώ ότι η σημαντική εστίαση θα πρέπει να είναι στο ότι θα καλύπτονται ακριβώς όλοι αυτοί οι τομείς. Κοιτώντας για παράδειγμα το share. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ο κόσμος που πάει διακοπές σε ένα ωραίο περιβάλλον με ωραίο καιρό αποτελεί μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα γιατί δεν είναι σε παγρύπνηση αν θέλετε. Άρα το κατά πόσον κάποιος είναι ευάλωτος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε με πιο ευρύ πρίσμα. Αντί να κοιτάξουμε, αν θέλετε, με ένα γενικό ορισμό για το επίπεδο απασχόλησης. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και τη βοήθεια της κυρίας Περές και ίσως να χρειάζεται και κάποια στατιστικά στοιχεία, μιας και έχουμε μαζί μας τον στατιστικό λόγο για πρώτη φορά έχουμε στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να ενταχθούν στη δουλειά της κυρίας Περές. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης, που είναι επίσης σκιώδης μετά την επιτυχία του την προηγούμενη εβδομάδα με την έκθεσή του, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Μάλκομ και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, γιατί εν πολύ συμφωνώ με αυτά που έχω ακούσει σήμερα. Συμφωνώ και μαζί σας κύριε Πρόεδρε ότι έρχεται αυτή η έκθεση στην καταλληλότερη στιγμή μετά την δική μου όπου έχω θίξει αυτή την έννοια του ευάλωτου καταναλωτή. Ε, συμφωνώ με την θέση που παίρνει η συγγήτρια ότι δεν πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή διότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάρα πολλοί από εμά μπορεί σε μια στιγμή να γίνουμε ευάλωτοι και την άλλη στιγμή να μην είμαστε. Ε, Ένα ορισμό που δίνεται συνήθω είναι ότι ο ευάλωτο καταναλωτή είναι ο μη επαρκώ ενήμερο καταναλωτή. Αλλά η ενημέρωση δεν είναι το παν για την ενδυνάμωση των καταναλωτών. Δεν τελειώνει δηλαδή η ενδυνάμωση του καταναλωτή με την ενημέρωση. Πρέπει να μιλήσουμε για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Για παράδειγμα, και το έθιξε η συγγήτρια ήδη, όπως το έθιξα και εγώ, τα μικρά παιδιά είναι πολύ ευάλωτα στην παραπλανητική διαφήμιση ε, λόγω του ότι δεν έχουν την ικανότητα, την οριμότητα, τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα άτομα τους από την διαφήμιση αυτή. Ε, όμως η παραπλανητική διαφήμιση δεν παραπλανεί μόνο μικρά παιδιά. Επίσης, η οικονομική κρίση στην, την οποία ε, διερχόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή νοθεί ανθρώπους να γίνουν πολύ πιο ευάλωτοι από ό,τι συνήθως θα ήταν. Επομένως, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το κράτος πρόνοιας και την κοινωνικότερη Ευρώπη όπου ο φτωχό, ο ανάπηρο, ο άρρωστο που δεν μπορεί να αγοράσει τα φάρμακα του, ο πεινασμένο να έχουν ουσιαστική βοήθεια. Και θα πρέπει να εισηγηθούμε τέλο αυστηρότερε ποινέ σε όσου κερδοσκοπούν σε βάρο των ευάλωτων, είτε αυτοί είναι άρρωστοι, άνεργοι, μικρά παιδιά κλπ. Επομένω, ε, θα αναμένω την έκθεση για να συνεργαστώ με την εισηγήτρια έτσι που να περάσουμε αυτά τα μηνύματα στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, and then Mrs. Head. Η κυρία Head. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω σου ειδικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία, όπως τη βλέπω, είναι πολύ επίκαιρη. Έχουμε σημαντική νομοθεσία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ε, ετών και συχνά έχουμε δώσει προτεραιότητα στις αγορές στα κείμενά μας. Οδηγία για τις υπηρεσίες, για την ασφάλεια των παιχνιδιών και άλλα σημαντικά θέματα όπου υπάρχουν ευαίσθητοι καταναλωτές και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία αυτή να, είναι, να ισχύει για όλους και να ταιριάζει σε όλους. Δεν πιστεύω πως όλοι οι καταναλωτές ε, γνωρίζουν τις ευθύνες τους. Μιλήσαμε για πολύ κόσμο που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος ε, για τους έφηβους, για τα παιδιά, τους ηλικιωμένου και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ε, θεωρηθούν υπεύθυνοι και γι' αυτό εμείς ως νομοθέτες πρέπει να σκεφτούμε την ε, περίπτωσή τους. Τα παιδιά, για παράδειγμα, πάντοτε μιλάμε για το θέμα της διαφήμιση που έχει μεγάλο αντίκτυπο στα παιδιά. Έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που χάρη σε αυτήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγαλύτερες ευθύνες στον τομέα αυτό. Είναι δουλειά μας να στηρίξουμε τα δικαιώματα των παιδιών και πέρα από αυτό τα παιδιά είναι διαρκώς εκτεθειμένα. Και ο εισηγητής είπε ότι είναι σημαντικό για μας να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν και αυτές ολόκληρη αυτή την προσπάθεια και την προοπτική, να συμμετέχουν ωστόσο και οι οργανώσεις των καταναλωτών, όπως και αυτές οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά. Οι, καταναλω... οι ενώσεις των καταναλωτών είναι αυτές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές και πώς μπορεί η κατάστασή τους να βελτιωθεί. Είμαι ευτυχής λοιπόν που είναι το θέμα στην ημερήσια διάταξη, που εργαζόμαστε από αυτού. Ελπίζω πως θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε όλους τους καταναλωτές να πάσα στιγμή στο μέλλον. Ξέρω το θέμα του ορισμού είναι δύσκολο, ε, αλλά και πάλι η νομοθέτηση είναι αυτή που θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τους καταναλωτές και κυρίως για τους πιο ευάλωτους εξ αυτών. Άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Τόμπρομ, θέλετε να μας πείτε ποια είναι η δικιά σας άποψη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα το κάνουμε ευχαρίστηση από την πλευρά της Κομισιόν και εμείς σε καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή. Πιστεύουμε πως είναι πολύ επίκαιρη γιατί θα είναι δυνατόν να συμβάλλει η έκθεση αυτή στη συνεχιζόμενη εργασία μας και στην προετοιμασία της επόμενης πολιτικής και στρατηγικής για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να πω επίσης πως η παρουσίαση της εισηγητρίας και ανάλυση της είναι πολύ σύμμορφη με τη δική μας, το δικό μας εσωτερικό προβληματισμό. Είναι δύσκολο βέβαια να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα των ευάλωτων καταναλωτών και όταν κανείς έχει ένα τεράστιο θέμα να αντιμετωπίσει, θα πρέπει να το τεμαχίσει σε μικρότερα κομμάτια. Και νομίζω πως αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος, γιατί θα δείτε πως η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την νομοθεσία αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και όταν εξετάζουμε τα υποκείμενα τα οποία υπόκεινται σε αυτή την νομοθεσία. Νομίζω πως η επόμενη ε, νομοθεσία θα είναι, και η εξέλιξη μάλλον αυτής θα είναι διαφορετική. Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να βρούμε ένα είδος ε, ένα επίπεδο που μπορούμε να συμφωνήσουμε, ποια θα πρέπει να είναι η προστασία των καταναλωτών, τι υπάρχει στα κράτη-μέλη. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα στην σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πράξουμε, να συζητήσουμε, γιατί μέχρι τώρα στο γενικό συμβατικό δίκαιο, ε, ενοχικό δίκαιο, αυτές οι ιδέες υπήρχαν και υπάρχει κάποια προστασία σε εθνικό επίπεδο συχνά τι είναι δίκαιο και ή άδικο σε μεμονωμένες ε, περιπτώσεις, συμβάσεις, αλλά επειδή το είχαμε αντιμετωπίσει και βρήκαμε λύσεις για τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει ωστόσο να δούμε το ενοχικό δίκαιο για τις διάφορες ε, νομοθεσίες. Γιατί στο μέλλον αυτό που μπορεί να λυθεί σε καταστάσεις προσωπικές μπορεί να ισχύει βέβαια, αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη και να λάβουμε υπόψη και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σίγουρα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να έχουμε μια κοινή ε, ε, βάση για το ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές υπάρχουν και είναι πολύ σημαντικό βασική ιδέα που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στην πολιτική μας για τον καταναλωτή. Η διασυνοριακή λοιπόν διάσταση καθιστά απαραίτητη την αντιμετώπιση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ γιατί επιβεβαιώσατε ότι συμφωνείτε και είστε στην ίδια γραμμή μαζί μας. Είναι ενδιαφέρον για τους συναδέλφους θα πρέπει να ορίσουμε τους, ε, με τους συντονιστές, αλλά έχουμε μία πρόταση επιτάπητος. Από ό,τι κατάλαβα η κυρία Τόμπλουμ ασχολείται με την πρόταση για μία κοινή δημόσια ακρόαση με τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για τους καταναλωτές. Προσωρινά το έχουμε θέσει για τις 19 Φεβρουαρίου. Τα αφήνουμε στους συντονιστές να συμφωνήσουν για αυτή την ημερομηνία. Αλλά αυτή είναι η πρόταση για την ώρα και φυσικά θα σας καλέσουμε να συμμετέχετε. Κυρία Ιρηγογέν Πέρες, θέλετε να ολοκληρώσετε πριν αρχίσετε να συντάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδης εισηγητές. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Μέσα σε αυτή την έκθεση δεν ε, επιχειρώ να εξετάσω την έννοια του ευάλωτου καταναλωτή. Περιγράφουμε μια κατάσταση επισφαλή. Δεν είναι μια στατική έννοια. Αντίθετα, είναι δυναμική, καθότι είναι αδύνατο να προβλέψουμε όλες τις επισφαλείς θέσεις οποίες μπορεί να περιέλθει ένας καταναλωτής. και όχι, δεν ε, Είχα καμία πρόθεση να μιλήσω για τους ευάλωτους καταναλωτές. Όπως είπαν οι σκιώδε. Ε, μιλώ για τον, την ευάλωτη κατάσταση των καταναλωτών. Για τα υπόλοιπα στοιχεία θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενημέρωση, οι οργανώσεις, οι ενώσεις καταναλωτών θα χρειαστεί να εμπλακούν πιο δραστήρια σε αυτήν την ε, ενημέρωση των καταναλωτών, να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στους καταναλωτές, κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς, όπου δεν είναι γνωστά κάποια στοιχεία, δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση. Ευχαριστώ πάντως ε, όλους τους σχεδόν ηγετές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Περιμένουμε με ανυπομονησία το πρώτο σχέδιο και φυσικά θέλουμε να δούμε και τις μελέτες και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά τα Χριστούγεννα. Θα περάσουμε στη δεύτερη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών. Καλωσορίζω και πάλι την κυρία Παρβάνοβα, την εισηγήτριά μας ε, σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Πολύ σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή. Θα σας δώσω το λόγο δεν έχουμε και πολλούς σκιώδεις εδώ από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πειράζει, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ασκατές εξελίξεις ε, στον τομέα της ε, αεροπορίες σχετικά με την ε, εμφάνιση αεροπορικών ε, εταιριών χαμηλού κόστους ε, κτλ. Δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τους επιβάτες και οργανώνουν τα ταξίδια τους αυτή η τελευταία με διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τομέας λοιπόν αφορά όλο ένα και περισσότερο τους καταναλωτές, αλλά πρέπει να κατοχυρώσουμε την κατάλληλη προστασία. Ε, ο κανονισμός 2061 το 2004 σε σχέση με τους κοινού κανόνες για την αποζημίωση των επιβατών και ο 1107 το 2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και με μειωμένης κινητικότητας συνέβαλαν στην σημαντική βελτίωση της κατάστασης. Παρόλα αυτά, δεν καλύπτονται ακόμη όλες οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιβάτες στα ταξίδια τους. Γι' αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ο 2006, το 2001 και ο 1107 το 2006 για να αντιμετωπίσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα. Δεν υπάρχει συνεκτικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου για τους επιβάτες ως προς τα δικαιώματά τους. Οι, οι ελλείψεις, οι ατέλειες, τη μεταγραφή στην εθνική νομοθεσία και στην ολοποίηση των νομοθετημάτων αυτών είναι ακόμη ένα πρόσκομα που μας απομακρύνει από την κατάλληλη προστασία των καταναλωτών οι νέες ρήτρες οδήγησαν σε περιπλοκές, σε διαφορετικέ ερμηνείε και οι καταναλωτέ δεν κατανοούν πλήρω τα δικαιώματά του. Χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τι έκτακτε περιστάσει. Αυτή για την έννοια των εκτάκτων περιστάσεων για να ενσωματώσουμε τι πρόσφατες αποφάσει του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των καταναλωτών υπό την επιφύλαξη τη ελευθερία των αεροπορικών εταιριών σχετικά με τι εμπορικέ του δραστηριότητε, θα πρέπει ε, τα τέλη για τις αποσκευές, ε, για το αυτοκίνητο αυτοκίνητο για την εγγραφή στο Μητρό Επιβατών να ληφθούν υπόψη ούτως ώστε να δούμε ποιο είναι το τελικό ε, ύψος ε, του αεροπαρικού ναύλου και αν είναι υποφελές ε, για τον καταναλωτή. Εσγάντω εγκρίθηκε και η οδηγία για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και θα πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην προστασία των επιβατών σε σχέση με την αεροπορική εταιρεία που κηρύσσει η πτώχευση ή που, της οποίας ανακαλείται η άδεια. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς επιλέγει ο καταναλωτής να αγοράσει το εισιτήριό του και να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα του αθέμητου ανταγωνισμού ανάμεσα σε αεροπορικές εταιρείες. Δεν ε, υπάρχει η πρόσφερη προς το παρόν διαδικασία για την αποζημίωση, την καταγγελία ε, από πλευράς των επιβατών και την αποζημίωση αυτών. Άρα προτείνουμε κατάλληλο συντονισμό σε σχέση με όλε τι νομοθεσίε που διέπουν τα δικαιώματα των επιβατών. Χρειάζονται επίση αναλλακτικά μέτρα για αναλλακτικέ διαδικασίε επίλυση διαφορών. Για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα, εκπονήσει η Επιτρο... θα έπρεπε η Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριε γραμμέ για την αναθεώρηση του κανονισμού 1107 του 2006 ε, για την ασφάλεια και για τα συνοδεύοντα άτομα, ώστε αυτά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν προστασία όταν δεν, τους, ε, δεν μπορούν να επιβιβαστούν λόγω της εταιρεία ή δεν διαθέτουν συνοδεύοντα άτομα. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που θα έπρεπε επίσης να ρυθμίσουμε στη μελλοντική ε, αναθεώρηση αυτών των δύο κανονισμών. Παραδείγματο χάρη, ε, αναλογικά αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπιση των αθέμητων όρων σύμβασης ε, ενοποίηση της νομοθεσίας ε, για αυτά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και για το χειρισμό των διαφόρων ε, μέσων που χρειάζονται για να μετακινηθούν. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ημερομηνία υποβολής τροπολογιών είναι σε 7 Δεκεμβρίου και στις 9 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση στην Επιτροπή Good. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Παρβάνοβα. Έχουμε το θέμα του μήκου ε, τη έκθεση. Είμαστε περιορισμένοι, αλλά σκιώδει συζητητέ ε, μα προσφέρουν προ τα αξία και αυτό ελπίζουμε. Ποιον έχουμε λοιπόν, η κυρία Τούν, ο κύριο Σαλβίν είναι εδώ από του σκιώδει. Κυρία Τούν, θα θέλατε να μα ε, παρουσιάσετε την άποψή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα ιδιαίτερα σε κάποιους μήνες του χρόνου όπου γίνονται τα πιο πολλά ταξίδια και θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα για τους επιβάτες είναι ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουν τίποτε. Έχουμε αυτή την φοβερή οδηγία για την οποία είμαστε τόσο περήφανοι και πολύ έντονα θυμάμαι τη μεγάλη επιτυχία θεωρήθηκε η υπερψήφιση της οδηγίας, αλλά πολύ συχνά μου δίδεται η εντύπωση ότι ούτε εφαρμόζεται, ούτε είναι γνωστή στον κόσμο. Και ένα από τα θέματα εδώ στην ε, έκθεση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει παντού πληροφόρηση για τα δικαιώματα των επιβατών. Κάποιες φορές σε κάποια αεροδρόμια βλέπουμε τέτοιες πληροφορίες, αλλά συνήθως βρίσκουμε πληροφορίες για το πού μπορεί να λάβει κανείς τις πληροφορίες. Ίσως θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει μια διαβούλευση για το πώς έχει ωφελήσει η οδηγία αυτή, κατά πόσον έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στα δικαιώματα των επιβατών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία. Άρα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε καταρχάς πολύ και πολλές πληροφορίες. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί και στη γνωμοδότηση. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο θεωρώ ότι λείπει στα αεροδρόμια, είναι ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός του τι σημαίνει τα συνοδεύοντα άτομα, άτομα με αναπηρία, τι ακριβώς περιλαμβάνουν, ε, το υπέρβαρο, τι, μάλλον άτομα υπέρβαρα, ποιοι περιλαμβάνονται και ποιοι όχι, πολλές ασάφειε. Η πρόσβαση στη βοήθεια. Ούτε αυτό ορίζεται με σαφήνεια. Λαμβάνει η βοήθεια όποιο το επιθυμεί, όποιο το χρειάζεται. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, δίδεται αυτή η βοήθεια, σε κάποιες άλλες τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία θα σα τα αναφέρω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλωστε, αλλά πολλές ε, πτυχές ε, εξελίσσονται, αν θέλετε, στα αεροδρόμια, τα οποία οι οποίες δεν αναφέρονται στην οδηγία. Για παράδειγμα, τα αεροδρόμια μετατρέπονται σιγά-σιγά σε εμπορικά κέντρα, με μαγαζιά. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη για το τι βάρος μπορεί κανείς να μεταφέρει καθαρά σε ψώνια στο αεροπλάνο γιατί συχνά ο κόσμος κάνει ψώνια και τελικά του επιτρέπεται μόνο μία βαλίτσα στο αεροπλάνο και τελικά δεν μπορεί να πάρει όλα τα πράγματα. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουν τα άτομα που δουλεύουν στα μαγαζιά σε ποια αεροδρόμια μπορούν να μεταφερθούν για παράδειγμα μπουκάλια, αλκοολούχα, ποτά. Δεν υπάρχει σχετική πληροφορία γιατί τα αγοράζει ο καταναλωτής σφραγισμένα και μετά δεν ξέρει πού μπορεί να τα, μεταφέρει, να, να τα μεταφέρει. Άρα, τα καταστήματα αυτά δεν είναι σωστά ενημερωμένα, ούτε θέλουν να ενημερώσουν τους επιβάτες για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αργότερα. Για πολλά προβλήματα θα περάσει, ελπίζουμε, το IDR η εναλλακτική επίλυση διαφορών θα έπρεπε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιείται πολύ πιο εντατικά για την επίλυση προβλημάτων μεταξύ επιβατών και αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών. Αυτά ως ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη εντύπωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας ε, παρουσιάζετε νέες ε, διαστάσεις. Ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά σας ε, για, το, για τα ψώνια μέχρι θανάτου σε οπτήλ τρόπο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι όντως υπάρχουν αβεβαιότητες. Και είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε στην πτυχή προστασία του καταναλωτή. Η κυρία Παρβάνοβα άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Πέρε, νομίζω ότι θα μιλήσετε εξ ονόματο των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Παρβάνοβα. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της. Συμφωνώ με τις γενικές ε, γραμμές ε, της επιχειρηματολογίας της εισηγήτριας. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ένα προβληματισμό. Υπάρχουν αλλαγέ ε, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Αυτό αληθεύει και είναι ταχύτερε από την εξέλιξη τη νομοθεσία μα. Θυμηθείτε τι έγινε με τον έφο σκόνη από το Ισλανδικό ηφαίστειο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομοθεσία στη νέα πραγματικότητα. Το άνοιγμα και η επέκταση του τομέα των αεροπορικών μεταφορών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση τη ποιότητα και περιορισμό των δικαιωμάτων των επιβατών, όπω είπατε. Χρειάζεται να προσφέρουμε στου καταναλωτέ ασφάλεια δικαίου. Τέσσερα είναι τα βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα ήδη το σχολιάσαμε. Θα πρέπει να προσέξουμε όλο ιδιαίτερο του ευάλωτου καταναλωτέ και πιο συγκεκριμένα τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, με κάποια αναπηρία. Ε, όπως και θεωρήσουμε τον τρέχοντα κανονισμό, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία των καταναλωτών. Δεν θα πρέπει, ξαναλέω, οι αλλαγές να μας οδηγήσουν σε περιορισμό των δικαιωμάτων. Τώρα, η ονομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως ως προς τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσει. Να καταπολεμήσουμε τον πολλαπλασιασμό των καταχρηστικών ερήτρων, παραδείγματο χάρη Επίση, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει να γνωρίζουν ναι, τα ένδικα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να είναι σωστά ενημερωμένοι. Ελπίζω να είναι καλό το τελικό αποτέλεσμα. Ε, μπορείτε να υπολογίσετε στη βοήθειά μου πάντως, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρούλ ε, θέλει το λόγο. Ποιος άλλος είναι εδώ? Ο κύριος Ντιγιό? Κύριε Σαλβίνη? Όχι. Ο κύριος Διγέων τότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη γιατί ίσως δεν ε, έχετε όλες τις εκθέσεις τις οποίες είμαι σκιώδης, θα το φροντίσω να το λάβετε. Θα ήθελα για την έκθεση αυτή να συμβάλλω ως σκιώδης. Πολλά έγιναν τον τελευταίο 1,5 χρόνο για... και πολλή αναστάτωση προκάλεσε το ηφαίστειο και πολλές ασάφειες ε, επικράτησαν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, σε ό,τι αφορά την ακύρωση πτήσεων στην Ολλανδία. Δεν ακολουθήθηκε δεν μπορούσε να ακολουθηθεί διαδικασία εθελούσιας επίλυσης γιατί αντιτάχθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες αλλά έγιναν τόσες πολλές καταγγελίες από επιβάτες που σε κάποια φάση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε να διευκρινίσει διάφορα ζητήματα και στην Ολλανδία μπορούν οι πολίτες να προσφύγουν στον δικαστή Μίλησα λοιπόν και με αεροπορικές εταιρείε και φαίνεται ότι θεωρούν ότι το, η τρέχουσα νομοθεσία ε, επιβαρύνει για οποιαδήποτε καταγγελία όλες τις αεροπορικές εταιρείε, ακόμα και για λόγους ε, που δεν ευθύνονται, δεν είναι στο πεδίο της ευθύνη των αεροπορικών εταιριών, ευθύνονται οι αεροπορικές εταιρείε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε στην ε, έκθεση. Και κατά δεύτερον, μία τάση σε κάποιες ε, αεροπορικές ε, εταιρείες να υποχρεώνουν άτομα υπέρβαρα να κλείνουν δύο θέσεις αντί για μία θέση. Νομίζω ότι αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και αποτελεί κάτι που είναι σε άμεση αντίθεση με αυτά που αποφασίζουμε για άτομα με αναπηρία, όπως είναι το υπέρβαρο τα υπέρβαρα άτομα. Νομίζω ότι θα πρέπει στο σημείο αυτό να τηρήσουμε τους υφιστάμενους κανόνες προκειμένου να γίνουν και κάποιες δευκρινήσεις και να μην τιμωρούνται από αεροπορικές εταιρείε τα άτομα τα υπέρβαρα. Πολύ μεγάλο έργο λοιπόν και φαντάζομαι ότι η συγγήτρια έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά και την περιορισμένη έκταση του κειμένου της γνωμοδότησης, αλλά και εγώ θα σας υποβάλω προτάσεις για να διασφαλιστεί και η πρόσβαση με ίσους όρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων αυτών των μέσων. Θεωρώ λοιπόν ότι έχετε πολύ μεγάλο έργο μπροστά σας. Good. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα παρουσιάσω κάποιες ε, απόψεις από την ομάδα μου. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τις νέες ε, διατάξεις όπως ανέφερε η κυρία Περμανοβά, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενισχυθεί το μήνυμα αυτό. Και σίγουρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση, γιατί αυτό έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή και έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ε, επιβατών και σε ό,τι αφορά την κράτηση εισιτηρίων Νομίζω ότι πολλά χρήσιμα στοιχεία ακούστηκαν για την προώθηση και την ενημέρωση ε, των επιβατών. Αυτό λοιπόν είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και για τα αεροδρόμια και για τις αεροπορικές εταιρείε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία έλλειψη συνοχής και κατανόησης σε ό,τι αφορά τα πραγματικά δικαιώματα των επιβατών. Ξέρω ότι έχουμε και δύο συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Ντίας Παλίτο. Θέλετε να πάρετε το λόγο, να σχολιάσετε στη φάση αυτή. Να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις, να σχολιάσετε προς την κυρία Παρβάνοβα, ίσως. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την προσπάθεια που έχει καταβάλει, για το χρόνο που έχει αφιερώσει στην ανακοίνωσή μας για τα δικαιώματα των επιβατών. Θα ήθελα να αναφερθώ στις πληροφορίες που αποτελούν ένα από τα αδύνατα σημεία, τα δυνάμα σημεία αν θέλετε. Το συνειδητοποιεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2009 ξεκίνησε μια έρευνα του Ευρωμαρόμετρου και ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τα δικαιώματα των επιβατών και έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δουλεύει. Εργάζεται επισταμένο ε, για τα θέματα αυτά. Ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ενημέρωση, την οποία και είδατε στις, ε, στα, στα αεροδρόμια. Όλε οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να κάνουν τέτοια ενημέρωση. Πέρσι ε, αποφασίσαμε να αντιοργανωθεί και μία ημέρα για τα δικαιώματα του επιβάτη και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σκοπεύουμε να τις επαναλάβουμε το 2012. Άρα, έχετε δίκιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία στην ενημέρωση και εργαζόμαστε από αυτού. Να πω ότι σημειώσαμε όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν και συμφωνούμε με την θέση της εισηγήτριας και της ε, πλειοψηφίας των βουλευτών θα περιμένουμε ίσως να δούμε και το τελικό κείμενο, το τελικό σχέδιο κειμένου για να κάνουμε περαιτέρω σχόλια, αλλά να σας πω ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν όλες αυτές οι ελλείψεις και συμφωνεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κρόιτσμαν δεν είχε λάβει το λόγο. Μία μικρή παρατήρηση Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε η συναδέλφο Τούν, ότι τα αεροδρόμια έχουν εγκαταστεί εμπορικά κέντρα. Και κάποιες φτηνές αεροπορικές εταιρείες για ένα επιπλέον πακέτο χρέων 40 ευρώ. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ενημερωθεί ο καταναλωτής. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να το πάρουν και αυτό υπόψη. Γιατί τελικά, αν δεν το ξέρει κανεί αυτό, αυτά που κλείτωσε στο duty free τα πληρώνει στην αεροπορική εταιρεία. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πρεβάνοβα, θέλετε ίσω να ολοκληρώσετε, να βγάλετε συμπεράσματα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να μας επιβεβαιώσετε και το τελικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε μέσω της έκθεσης αυτής, γιατί όλοι μας έχουμε πέσει θύματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μιας και ταξιδεύουμε τόσο συχνά. Όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία της έκθεσης αυτής στο γραφείο μου, λάβαμε πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλές πληροφορίες από ενώσεις καταναλωτών και από αεροπορικές εταιρείες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια σύνοψη η οποία και να χωρέσει μετά σε μια μικρή γνωμοδότηση. Γι' αυτό νομίζω ότι για το μέλλον ο τομέας αυτός τι να σας πω, θεωρώ ότι έχει περιθώριο για πλήρη έκθεση από πλευράς της ΙΜΚΟ σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τώρα, δεδομένων των περιορισμών, θα ήθελα να προτείνω στους συναδέλφους να καταθέσουν κάποιες ε, τροπολογίες, γιατί υπάρχουν τόσο πολλά θέματα, τόσο πολλά ζητήματα, τα οποία δεν θα είμαστε σε θέση να τα χωρέσουμε στην ε, γνωμοδότηση προς την Ήτρε. Άρα μπορούμε να καταθέσουμε με τους κοιόδες κατευθείαν τις ε, τροπολογίες αυτές στην Επιτροπή Ήτρε. Ο Πρόεδρος. Α, ναι, ίσως τις μεταφορές ε, εννοούσατε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές η σχέση μας ε, με την Επιτροπή Μεταφορών και νομίζω ότι θα δεχτούν να λάβουν τροπολογίες από άλλες επιτροπές. Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο και θα περιμένω και τις συστάσεις σας για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα γίνει στην ε, Επιτροπή Μεταφορών η ψηφοφορία για την τελική έκθεση. 9 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα με την ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ. Προφανώς ε, μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες και στην Επιτροπή Μεταφορών. Αν θα θέλατε να το ενθαρρύνετε αυτό θα ήταν θετικό θεωρώ. Ωραία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Είναι περασμένε 10. Θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίε. Δεν είμαι βέβαιο αν έχουν έρθει όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 10 η ώρα είχαμε πει. Άρα θα ξεκινήσουμε τι ψηφοφορίε. Και έχουμε και αρκετέ σήμερα. Καταρχά, έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση τη Σαλβίνη και τον εξυγχρονισμό των τελωνίων μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, 110 τροπολογίες. Νομίζω, μιας και δεν είχαν γίνει πάρα πολύ εκτενεί συζητήσει για τις τροπολογίες, μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα λίγο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σαλβίνη. Σας παρακαλώ μόνο λίγη ησυχία για να συζητήσουμε. Κύριε Σαλβίνη, Θέλετε να πείτε δύο λόγια πριν την ψηφοφορία και αν θέλουν κάποιοι σκιώτες να πάρουν το λόγο θα τους δώσω λίγο χρόνο. Αλλά καταρχάς ο λόγος των εισηγητή. Grazie Presidente, ringrazio lei uffici e tutti i relatori ombra per il prezioso ε, Ευχαριστώ καταρχήν τους κοιόδης ηγητές για την πολύτιμη του συμβολή. Καταφέραμε 11 συμβαστικές ε, τροπολογίες που σημαίνει Πολύ δουλειά εις βάθος. Υπάρχει και η ένδειξη μιας ενημερωμένης ημερομηνία που ευχόμαστε να εγκριθεί και την υποβάλλουμε στην Κομισιόν ως νέο στόχο για την έναρξη ισχύους του ανανεωμένου τελωνιακού κώδικα. Ελπίζω να μην υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές σε αποχρώσεις και σε οπτικές για ορισμένε λεπτομέρειες για τους έλεγχους που θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί σε σχέση με εμπορεύματα που προέρχονται από ορισμένε χώρες και όχι σε σχέση με τις ε, ενδείξεις, υποδείξεις που θα πρέπει να κάνουμε στις άλλες επιτροπές. Πιστεύουμε ωστόσο πως το κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές ε, λαβές για την νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία εφόσον στις συνεδριάσεις της, ε, των προηγούμενων εβδομάδων ε, δεν είχαμε αντιμετωπίσει όλα τα κύρια θέματα συζήτησης και τα έχουμε λύσει βασικά με τις 11 συμβιβαστικές, επί δύο επί ε, εκ των οποίων δύο έχει συζητηθεί τμήματική ψηφοφορία, αλλά πάντως το μεγαλύτερο τμήμα της δουλειάς έχει γίνει χάρη στην προσήλωση όλων. Σας ευχαριστούμε πολύ που καθοδηγήσατε όλη αυτή τη διαδικασία και νομίζω πως έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση εδώ και πάλι επίκαιρη. Η κυρία Ράπτη που είναι σκιώδης εισηγήτρια από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σαλβίνη για τη δουλειά που έκανε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους Σκιώδης, καθώς εργαστήκαμε όλοι μαζί σε μια πολύ καλή βάση, πάνω σε ένα πολύ καλό κείμενο που έκανε ο κύριος Σαλβίνη. Θεωρώ υποχρέωσή μου να το υπογραμμίσω, γιατί νομίζω ότι ε, η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι προς το να βρίσκει τους καλύτερους δυνατούς συμβιβασμούς σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για την ευρώπη προκειμένου να ωφελούνται οι ευρωπαίοι πολίτες. ευχαριστώ και πάλι ήταν μια ε, πολύ χρήσιμη εμπειρία για μένα αυτή η συνεργασία και αυτή η έκθεση. ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much for that. Uh, I'm sure Mr. Σας ευχαριστούμε. Σίγουρα ο κύριος Σαλβίνη θα το σκεφτεί πολύ, γιατί είναι η πρώτη εκθέση που συντάσσει για την Επιτροπή μας. Υπάρχει κανένα άλλο που θα ήθελε το λόγο. Όχι, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία αν χρειαστεί. Έχετε τι κάρτε, αλλά προ το παρόν δεν νομίζω ότι χρειάζεται επαλήθευση. Τελό πάντων, να προσπέχουμε τα νούμερα. Α αρχίσουμε με τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Ε, σαφέστατα εγκρίνεται. 15 τώρα. Κύριο Πάτσα, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τώρα, 21. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. 24 υπέρ. Κατά επίσης εγκρίνεται. 25 καταπίπτει. 26 τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. Ίντα ένα. Είναι όλα αντίστοιχα μέρη. Corresponding parts. Ε, δεν θα τα δούμε μονομένα, απλώ για να καταλάβετε που είμαστε στον κατάλογο ψηφοφορία. Ε, είναι τα ένα υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Είναι τρία. Και το αντίστοιχο τμήμα υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. 27 της κυρίας Ρούλε τώρα. Υπέρ. Κατά. Σαφέστατα απορρίπτεται. 28. Κύριε Σκόχαλε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Υιοθετήθηκε. 36 τώρα της κυρίας Δουρολέ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Είναι τα πέντε. Επίσης αντίστοιχο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 τώρα. Του κυρίου Σμιτ και άλλων υπέρ. Νομίζω χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 35 παρακαλώ. Πέρας. 16 προς 16, άρα απορρίπτεται. 37 του κυρίου Ντιγιόν υπέρ κατά. Α, απορρίφθηκε. 38 υπέρ. Επαλήθευση παρακαλώ για την 38 του κυρίου Ντιγιόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται η ισοψηφία 16 προς 16. 30 της κυρίας Κόχολα υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41. Η 40 έχει εγκριθεί, όπως λέγαμε, και λέει ο κατάλογος ότι υπάρχουν κάποιες πρόσθετες λέξεις για τη 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 42 του κυρίου Ντιγιόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Τώρα. Είναι τα 6 Σωστά τα λέω, ναι. Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, τροπολογία 6, αντίστοιχο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 52 της κυρίας Δράπτη. Ηλεκτρονική παρακαλώ, για την 52. Πέρας. Ε, εγκρίθηκε με 21 υπέρ 11 κατά. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Είναι τα 5. Το αντίστοιχο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 57. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 τώρα είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία που ζήτησαν δύο πολιτικές ομάδες. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ, βλέπετε στον κατάλογο σας, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε με 18 προς 15. τώρα. 64, αν δεν κάνω λάθος, ένα λεπτό. Είναι λίγες σελίδες μετά. Τι του κύριο Ντιγιό, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 7, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 8, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 9, το αντίστοιχο τμήμα. Κατά, Επίσης εγκρίνεται. Τώρα επί, ε, πρόσθετες λέξεις κυρίας Κόχολα για την 65 υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Τώρα, 66 έχει αποσυρθεί. 67 του κυρίου Σφάμπ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται και τώρα 73 υπέρ κατά εγκρίνεται 74 74 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας Εγκρίθηκε με 20 προς 13 ψήφους. 78 τώρα. Το αντίστοιχο τμήμα, corresponding part, ο κύριο Σμιτ και άλλων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 20 προς 13 ψήφους. Νομίζω ότι είναι τα δύο καταπίπτει. Η 75 επίσης καταπίπτει. Άρα πάμε στο δεύτερο τμήμα της 75 του κυρίου Σφάμπ. Άρχεται. Για το 75 αντίστοιχο τμήμα 2 του κυρίου Σφάμπ. Πέρας. 20 προς 12 εγκρίνεται. 78 τώρα, το αντίστοιχο τμήμα 2. Πρόκειται για την ε, τροπολογία για την παράγραφο 16 πέρα Α, ηλεκτρονική επαλήθευση είναι ευχερέστερο. Για την 78 παρακαλώ. Το αντίστοιχο τμήμα 2 για την παράγραφο 16 πέρας εγκρίθηκε με 20 προς 13 ψήφους. Πού πάμε τώρα? Είναι τα δύο καταπίπτει, αν δεν κάνω λάθος. Το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα, λοιπόν, θα ψηφίσουμε τις ίντα 2. Με ένα αντίστοιχο τμήμα. Παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε με 20 προς 13 ψήφους. Η 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 77 τώρα. Άρχεται. Πέρας. Απεριφθεί. Σαφέστατα. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Ε, η ένα της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών η 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τη ίδια Επιτροπή η 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. τα 4. Το αντίστοιχο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 4, το αντίστοιχο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επιτροπή Ελέγχου 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επιτροπή Ελέγχου 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Της Ιδίας Επιτροπής 9 υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. Η 86 του κυρίου Σφαμπ. Νομίζω η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι καλύτερα. Η 86 παρακαλώ. Πέρασε. Κάποιος αργεί. 18 προς 12. Είναι ψήφι εγκρίνεται. 22, ε, παράγραφος 22, 87 ε, και 88 ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ. Κατά. Α, σαφώς απορρίπτονται. Η 89 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται αναμφίβολα. Τώρα θα περάσουμε στην 90 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Ε, ε η 91 του κύριου Έγκστρομ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 93 το πρόσθετο τμήμα, τα πρόσθετα τμήματα υπέρ κατά εγκρίνονται. Η 94 υπέρ κατά εγκρίνεται. 95 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται με 21 ψήφους προς 12. Η 96 τώρα παρακαλώ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 97 καταπίπτει λοιπόν. 98 της κυρίας Δράπτη υπέρ κατά εγκρίνεται. 99 καταπίπτει και η 100. Καλά τα λέω. 101 υπέρ κατά εγκρίνεται. Είναι τα 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 109 του εισηγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Είναι τα 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Είναι τα 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντα. 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 3 είναι ένα πρόσθετο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Επίση 9 υπέρ κατά Επίση εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται Κατά ήσασταν εσεί? Ε, είμαι πολύ γρήγορο. Ένα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνουμε όλες τις τροπολογίες. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Παρακαλώ ψηφίστε για το σύνολο της έκθεσης. Πέρας. Εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, καμία, κατά καμία αποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαλβίν. εξαιρετική η έκθεσή σας. Um, I think, um, I think it's Εγκρίναμε πολυπληθείς τροπολογίες και από τις ε, δύο επιτροπές διεθνούς εμπορίου, δηλαδή και ελέγχου τον προϋπολογισμό. Αυτό βοηθάει, όπως ξέρετε, γιατί συχνά συζητιέται αυτό το θέμα των εργασιακών μας ε, σχέσεων και της συνεργασίας μας με άλλες επιτροπές. Ο κύριος Σαλβίνη μπορεί να στείλει μια επιστολή στους Προέδρους των δύο επιτροπών για να τους ε, ευχαριστήσει για τη συμβολή τους. Δεν ε, συνηθίζεται, αλλά νομίζω ότι καλό είναι για να υπάρχουν αγαστές σχέσεις και προσφέρει επίσης υποστήριξη και για την έκθεση. Επίση χρειαζόμαστε κατάλληλο χρόνο αγόρευση για τον εισηγητή. Συγγνώμη, αλλά ένα λεπτό για τον εισηγητή. Για τόσο σημαντικέ εκθέσει ε, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση και πρέπει να πηχείται και ο όγκο ε, τη δουλειά των εισηγητών. Αν λοιπόν συμφωνεί η Επιτροπή θα ζητήσω ε, περισσότερο χρόνο αγορός. Πολύ ωραία. Περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο, την έκθεση του κυρίου Μπίλαν. Είναι μία ε, γνωμοδότηση για προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για το Γραφείο Εναρμόνων στο πλαίσιο τη αγοράς αγορά ε, και αναθεώρηση της εντολής του. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπίλαν για να κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση πριν την ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους κοιόδης εισηγητές και το προσωπικό της γραμματείας και την κυρία Γιούλια Φαρνάιτ κυρίως. Εργαστήκαμε ταχύτατα για την εκπόνηση της ε, γνωμοδότησης για να ολοκληρωθεί η Επιπολωνικής Προεδρίας χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που χάρη στους ε, συναδέλφους μου από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ε, επιτύχαμε το στόχο μας. Καταλήξαμε σε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες και πρωτού καν αρχίσουμε την ψηφοφορία θα ήθελα να σας πω ότι υπέβαλα και μία προφορική τροπολογία γιατί μου το ζητήσαν πολλοί σκιώδεις εισηγητές. Πρόκειται για το άρθρο 4, είναι η τροπολογία 10 και προσθέτουμε εκεί ενώ τηρούμε το απόρριτο κτλ. Ελπίζω με αυτή την προσθήκη θα επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ε, είναι όντως σημαντική η γνωμοδότηση αυτή και χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε και εμείς για αυτή την πρόταση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27. Μπάστος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28, όπου έχουμε τμήματική ψηφοφορία που έχει ζητηθεί από το ΕΛΚ. Θα ψηφίσουμε πρώτα για το τμήμα 1 της τροπολογίας 28. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18 προς 14. Τώρα, εδώ δεν χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Υπέρ της πρώτου δεύτερου τμήματος, κατά, απορρίπτεται. Σαφώς. Περνάμε στην τροπολογία 4. 4. Ψηφίζουμε για την 4. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ 10 κατά και εφόσον εγκρίθηκε ψηφίζουμε η τροπολογία 29 της κυρίας Βερνιέ ως ε, επιπλέον σημείο υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 30 που αν υιοθετηθεί θα αναδιατυπωθεί υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά εγκρίνεται και τροπολογία 32 προσθήκη αυτών των λέξεων υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 34 Βαν... Βερνιό, υπέρ. Πέρας ψηφοφορίες. απορρίπτεται με μία ψήφο 16 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 35 Βερνιό, ποια είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 36, να ψηφίσουμε. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Κύριε Μάγερ, δεν τα καταφέρατε. Οι 37 και 38 έχουν αποσυρθεί. Πάμε τώρα στη ε, τροπολογία 9 του εισηγητή περ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Εδώ έχει ζητήσει το ΕΛΚ τμηματική ψηφοφορία. Οπότε ας ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα πρώτα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Για το τμήμα 2 Ας ψηφίσουμε για το 2, το δεύτερο τμήμα μάλλον, τέλος της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 17 ψήφοι κατά και 15 υπέρ. Προχωράμε στην 10 με την προφορική τροπολογία που ήθελε να ψηφίσουμε ο κύριος Βίλαντ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 τώρα, υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 44 καταπίπτει, 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 45 και 46 υπέρ κατά εγκρίνονται. Συμβιβαστική 2 ποιοι είναι υπέρ κατά εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 3 ποιοι είναι υπέρ κατά εγκρίνεται και τροπολογία 18 μπάστος με την προφορική τροπολογία που βλέπετε ποιοι είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται τροπολογία 19 προφορική της κυρίας Μπάστος ψηφίζουμε για τη 19 τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τώρα να ψηφίσουμε για τη 19 χωρίς την προφορική. Μάλιστα. Ψηφίζουμε για τη 19 χωρίς την προφορική τροπολογία. Vote is closed. And that's also... Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Πάμε στην 2, όπου ο κύριος Μπίλαν υπέρ, υπέρ κατά εγκρίνεται. Επιπλέον ε, προσθήκη λέξεων στην τροπολογία 20, υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 21, μπάστος, υπάρχει εδώ έτοιμα για κατατμήματα ψηφοφορία. Το έχει ζητήσει η ομάδα των σοσιαλιστών. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και για το δεύτερο τμήμα τώρα, ηλεκτρονικά. Closed. And that's rejected. Uh, so we now move to. Τροπολογία 22 τώρα. 22 ποιοι είναι υπέρ. Ε, έχουμε, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Και εδώ έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Uh, we Uh, um, final Και φτάνουμε έτσι στην τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λοιπόν αρχίζει τώρα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. As Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται χαλαρά. Κανείς δεν είναι κατά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίλαν. So we hope that you will be able to defend our amendments with the Legal Affairs Committee. Ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τις τροπολογίες νομικής επιτροπής και περνάμε σε μια άλλη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την Ευρώπη και την Κίνα. Εμπορική ανισορροπία και ερωτηματικό ανισορροπία. Ο εισηγητής δεν είναι εδώ, δεν νομίζω. Αν ο κύριος Κούρσμα θέλει να μας πει κάτι, εξ ονόματος του κυρίου Λεκεγκάρντ. Ναι, θα ήθελα να πω ε, τον κύριο Λεκεγκάρντ, ο εισηγητής θα ήθελα να απορρίψει ε, ε, το αίτημα για τη συμβαστική 5 σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα αυτή που θεωρεί ότι είναι αντιπαραγωγική. Αυτή είναι η μοναδική παρατηρήση που θέλω να κάνω. Ωραία, λοιπόν, θα το κοιτάξουμε όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Αλλά προφανώς, αν είναι αντίθετο σε προφορική τροπολογία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Let's... Μάλιστα, προχωρήσουμε λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη. Να περάσουμε πάλι στην ε, τροπολογία 8 της κυρίας Μακλάρκη. Τροπολογία 8. 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη 17 τώρα. Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Η προφορική τροπολογία για την 5 ε, δεν έχει τη συμφωνία μιας πολιτικής ομάδας, άρα δεν την δεχόμαστε. Και τώρα περνάμε στην 6, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Περνάμε στη συμβαστική 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 5 υπέρ. Να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Ηλεκτρονικά. Uh, the vote is closed. Uh, and that's... Τέλος. Α, απορρίπτεται. Δύο δεν ψήφισαν. Δεν είσαστε αρκετά γρήγοροι. Η 43. Έναρξη ψηφοφορία. Have 33 so that's closed. And that's rejected by... Απορρίπτεται. Η 44 της κυρίας Μακλάρκιν. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. The uh, vote's closed. And that's carried by 21. Πέρασε, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου ε, γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Uh, the vote's closed. And that's carried by 28. Πέρας ψηφοφορία, 28 ψήφοι υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λόικεγκάρτ να του μεταβιβάσετε τα συγχαρητήρια, κύριε Κρόιτσμαν. Και τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν για την ενοποίηση και την ε, εξέλιξη της διαδικασίας της Μπολόνια, ε, Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Σχετίζεται με το έργο της κυρίας Μακλάρκιν. Δεν ξέρω, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Αυτό εντάσσεται στο έργο που κάναμε στην Επιτροπή για τις επαγγελματικές δεξιότητες. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί η διαδικασία της Μπολόνια σε ό,τι αφορά την διατύπωση και τον ορισμό ε, των δεξιοτήτων και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων. Και άκουσα επίσης ότι στην Επιτροπή θα λάβουν υπόψη τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σε μεβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 10 υπέρ για την 10 ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Έναρξη ψηφοφορία για την 12. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 7. Έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Το έχουν ζητήσει οι πράσινοι. Δύο τμήματα λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 2 υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται κενό και τώρα νομίζω ότι περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Ένας δεν έχει ψηφίσει. Λείπει μία ψήφος. Μάλιστα. Εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν και πάλι είναι πολύ καλή, ήταν πολύ καλή η δουλειά σας. Είσαστε μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού είσαστε σε πάρα πολύ καλή θέση να προασπίσετε τις θέσεις και τις τροπολογίες της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά το τελικό έργο της Επιτροπής Πολιτισμού. Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα ο κύριος Πιτέλα ε, έλπιζα ότι θα είχε καταφτάσει, αλλά σε 10 λεπτά θα έρθει. Μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς τον κύριο Πιτέλα. Μας ε, είπε ο κύριος Πιτέλα ότι θα έρθει στις 11 παρα 5. Αλλά δεν θέλω να περιμένουμε. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να αναλάβει την ψηφοφορία εξ ονόματος του κυρίου Πιτέλα. Η ε, κυρία Κέπχαρτ ναι, Πρόεδρε, εγώ προτείνω να περιμένουμε για τις... Ε, μάλλον σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχουν αφιλεγόμενα ζητήματα. Ο κύριος Πιτέλα είναι ευγνώμων για την καλή συνεργασία, αλλά νομίζω να ψηφίσουμε, να μην κάνουμε διάλειμμα 10 λεπτά. Εγώ θα προσπαθήσω να το διευκρινίσω και να το εξηγήσω και στον κύριο Πιτέλα. All well, thank you very Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Νομίζω ότι πολύ καλή δουλειά έκανε. Να ψηφίσουμε. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Για μια ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά. Για την... Ε, καταρχάς, ε, τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ως προσθήκη και αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά για την 6. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Χαίρομαι που συμμετέχουν πιο πολλοί συνάδελφοι στις ψηφοφορίες. Εφτάσαμε τους 35. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία. 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 8. Ένταξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία 3 ως προστίκη. Η τροπολογία 3 ως προστίκη. Έναρξη ψηφοφορία Η τροπολογία 3. Πέρασε. 17 υπέρ, 17 κατά, άρα απορρίπτεται. Ο ένας που δεν ψήφισε θα ήταν ε, καθοριστική σημασία. Όπως και να έχει απορρίφθηκε. Και περνάμε στο 15 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 28 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 13 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Και χαίρομαι που ήρθε και ο εισηγητής μα, ο κ. Πιτέλα. Καλώς ορίσατε. Ξεκινήσαμε χωρίς εσάς. Τουλάχιστον θα μου θα ψηφίσετε ένα τμήμα τη έκθεση. Η 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 ω προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 20 καταπίπτει. Η 9. Σε τμήματα. Για την 9. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 23 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 22. Καταπίπτει. Α, όχι. 22, 22, υπέρ. Ω προσθήκη. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 26 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 25 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Η 13. Η 30, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 10 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και η 31 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πριν ψηφίσουμε, χαίρομαι που ήρθε ο εισηγητής και θα του δώσω λίγο το λόγο. Αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο πριν την τελική ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ συγγνώμη που ήρθα λίγο καθυστερημένα. Εσεί ε, τελειώσατε πιο γρήγορα, ε, περίμενα να είναι λίγο αργότερα. Ήμουνα σε μια διάσκεψη τη Επιτροπής ε, της Οικονομικής και της Κοινωνικής, γι' αυτό άργησα. Σας ευχαριστώ πολύ για την θετική υποδοχή που είχε η έκθεσή μου. Εξάλλου προσπάθησα να ε, δεχτώ σχεδόν όλες τις τροπολογίες γιατί ήταν θετικές οι προτάσεις που περιλάμβαναν. Είναι μια γνωμοδότηση την οποία συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Good. Well, let's Πολύ ωραία, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. είμαστε, 36 που ψηφίζουμε. Κύριε Πιτέλα, οι περισσότεροι ψηφοφόροι για σήμερα. Τρεις έχουν βάλει τις κάρτες αλλά δεν ψήφισαν. Όχι. Ορισμένοι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Εντάξει. Αλλά είναι ένας παραπάνω. Ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Κύριε Πιτέλα, μην ψηφίζετε υπέρ της έκθεσής σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα. Ο συντονιστή σα έδωσε το ψήφο του. Μα τι γίνεται, φεύγουν όλοι. Τέλος ψηφοφορίες. 33 ψήφισαν, 33 υπέρ. Κανείς δεν είναι κατά. Μπράβο, κύριε Πιτέλα, ευχαριστούμε. Έτσι τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Ε, η παρουσίαση της κυρίας Γκέπχαρτ θα ξεκινήσει στις 11. Η Κομισιόν δεν είναι ακόμα εδώ, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 11, αν συμφωνείτε. Διάλειμμα μέχρι τις 11.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

βέβαια Okay, ladies and gentlemen, I think we'll. Um, like to um, now to um, resume the. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με το τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί. Πρόκειται για την ε, εργασίε μα στο έγγραφο εργασία σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών. Ε, πριν ε, καλέσω την εισηγήτρια μα παρουσίαση στο έγγραφο, θα ήθελα να σα ενημερώσω για δύο εξελίξει. Πρώτον, Συνεχίζουμε συζητήσει με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με το ποιος, ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια κατά κύριο λόγο για αυτή την έκθεση. Ούτω ή άλλω θα υπάρξει στενή συνεργασία, όποια κοινή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θέτει εν αμφιβόλο την ε, αναπομπή της έκθεσης και άρα η διάσκεψη των Προέδρων θα πρέπει να αποφασίσει. Εμείς προετοιμάζουμε τη θέση μας, είναι ισχυρή τώρα, την οριστικοποιούμε και θα πάει στον κύριο Λένε σήμερα, στον πρόεδρο της διάσκεψης των Προέδρων δηλαδή, για να συνηγορήσει υπέρ της Επιτροπής μας. Ε, θα πρέπει να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά αυτή την υπόθεση μέσα από αυτή τη θέση μας. Η κυρία Γκέπχαρτ να αναφέρω επίσης ότι ε, συναντήθηκε με το διοριστέτη εισηγητή από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Τον προσκαλέσαμε φυσικά να παρευρεθεί στην ε, σημερινή συνεδρία, δεν τον βλέπω όμως. Ανήκει στην Γκουέν, ο κύριος Κλούτα συνάδελφος του κ. Ντιγιόν. Ε, έχουμε και μία μελέτη από την, ε, το Τμήμα Πολιτικών για τις ε, Τραπεζικές Υπηρεσίες. Έχετε λάβει αντίτυπο. Δεν προλάβαμε να τη διαβάσουμε, αλλά νομίζω ότι η πρόταση έγινε στο εξή. οι συντάκτες από το LSE θα έρθουν τον Ιανουάριο για να μας παρουσιάσουν τη μελέτη και έτσι θα συνεχίσουμε εμείς τις εργασίες μας. Ε, συλλέγουμε υλικό για το θέμα πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτά που μας έχει δώσει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, παρότι έχουν ήδη οργανώσει ακρόαση και νομίζω ότι η κυρία Γκέπχαρτ ήταν εκεί. αυτή, έτσι έχει η κατάσταση, αν θέλετε, προς το παρόν. Δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε από το να εξετάσουμε εντελεχώς το ζήτημα, διότι η κυρία Γκέπχαρτ ούτως ή άλλως έχει εργαστεί άοκνα. Παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Κατόπιν θα ακούσουμε τους Κιώδης, ο κύριος Μάγιος, ο κύριος Κρόιτσμαν, εξ ονόματος του κύριου Σμιτ, αν δεν κάνω λάθος, και η κυρία Τούρινεν, ε, αντί του κύριου Κέμφερ, ο κύριος Φόξ απουσιάζει, αλλά έχω τις σημειώσεις του, ο κύριος Ντιγιόν είναι εδώ. Οπότε έχουμε αρκετού σκιώδει συζητητέ. Κύριε Γκέπχαρτ, ε, θα σας δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσετε το έγγραφο εργασία σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι με πολύ πετυχημένο τρόπο περιγράψατε τη διαφωνία μεταξύ των δύο επιτροπών. Όντω, ε, θεωρώ ότι το θέμα είναι μια παρεξήγηση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ η έκθεση πρωτοβουλίας αυτή για τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αποτελεί το στόχο του κειμένου αυτού. Η Επιτροπή Οίκων έχει κατά νου ότι προφανώς υπάρχει κάποια υποχρέωση να δοθεί σε κάθε πολίτη πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ανεξάρτητα από την τράπεζα. Αυτό ωστόσο δεν το λέει η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, το θέμα είναι το δικαίωμα του πολίτη να μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό. Στη σημερινή εποχή που πολλά συμβαίνουν μέσω ίντερνετ, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, που πολλά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τραπεζικό λογαριασμό. Εδώ μιλάμε για προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες να λαμβάνουν όντως την πρόσβαση αυτή και είναι στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να ορίσουν με ποιο τρόπο θα το πετύχουν αυτό, με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Αν θα υποχρεωθεί μία τράπεζα, πολλές, όλες οι τράπεζες να προβούν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Αυτά περιλαμβάνονται και επαφίονται στα κράτη-μέλη στην πρόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε που διορίστηκα εισηγήτρια ασχολήθηκα εντελεχώς με το θέμα και πρέπει να ομολογήσω ότι αναγκάστηκα να ξεπεράσω και κάποιες δικές μου προκαταλήψεις και κάθισα και σκέφτηκα ποιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιαστικά. Τα άτομα με πιο περιορισμένα μέσα, αυτά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση για να συμμετάσχουν στην κοινωνία. Και όντω ε, πρόκειται για αυτά τα άτομα σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που είναι διαφορετικές. Πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Με πολλούς τρόπους. Στην Κρακοβία, όταν συμμετείχαμε στο φόρουμ για την ιστορική αγορά, αντιμετωπίσαμε και μια συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία θέλω να σας περιγράψω. Μια νεαρή φοιτήτρια η οποία είχε λάβει υποτροφή Εράσμου σε μια χώρα, ήθελε να συνάψει σύμβαση εκμίσθωσης. Τη ανέφεραν όμως, κοιτάξτε, στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν χωρί τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα μας να μισθώσετε κάτι. Μάλιστα να ανοίξει λογαριασμό, είπε. Ήθελε να ανοίξει λογαριασμό, λοιπόν. Αλλά στην τράπεζα τη είπαν, κοιτάξτε, λυπούμαστε, αλλά δεν μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό όσο δεν έχετε διεύθυνση στη χώρα. Και τώρα αυτό αποτέλεσε πραγματικό πρόβλημα για την νεαρή γυναίκα η οποία ήθελε να ζήσει στην Ευρώπη και αντιμετώπισε πρόβλημα. Δεν είχε πρόσβαση στην τράπεζα με τρόπο τελείως ακατανόητο. Στο πολύ ενδιαφέρον έγγραφο του, της υπηρεσίας κατάστροφης και σχετικής πολιτικής βλέπουμε και άλλα ενδιαφέροντα παραδείγματα όπως για παράδειγμα ότι στο Λουξεμβούργο το να μην μιλάει κανείς τη γλώσσα μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης για το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Και πολλά άλλα παραδείγματα μπορούμε να παρουσιάσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι να δώσουμε στους πολίτες να κινούνται όντω ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην αποτελεί πρόβλημα το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε μια χώρα στην οποία διαμένουν, ε, φοιτούν, δουλεύουν. και τελικά να μην έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και μετά να αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες επειδή δεν έχουν ακριβώς λογαριασμό στη χώρα αυτή. Ένα άλλο θέμα το οποίο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλήσαμε και για φοιτητέ οι οποίοι δεν έχουν κατά κανόνα πάρα πολλά χρήματα. Είναι το πόσο υψηλά επιτρέπεται να είναι τα τραπεζικά τέλη για τη λειτουργία ενός λογαριασμού. Θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να είναι δωρεάν. Αυτό δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρύνονται υπερβολικά. Τέτοια λοιπόν ζητήματα επεξεργαζόμαστε και επιχειρούμε να ορίσουμε στο πλαίσιο αυτό. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα βασικό λογαριασμό. Έναν λογαριασμό με τον οποίο μπορεί κανείς να, να διεξάγει τις γενικές υπηρεσίες. Δεν προβλέπεται η παροχή όλων των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η αγορά μετοχών κτλ. Όχι, έναν βασικό λογαριασμό. Αυτό αποτελεί το αντικείμενο ε, για να έχει κανείς ελευθερία κίνησης, να έχει πρόσβαση στα χρήματά του και αυτό αποτελεί ένα θέμα πολύ σημαντικό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και για μας, πάντα ήταν άλλο σημαντικό στην Επιτροπή μας, είναι το πώς μπορεί κανείς να απαιτεί στα δικαιώματά του όταν υπάρχει πρόβλημα σε μια τράπεζα για το άνοιγμα ενός λογαριασμού και άρα η παράγραφος όπου εξετάζονται τα ζητήματα της συλλογική ε, καταγγελίας ή της ε, επίλυσης διαφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική αυτή η παράγραφος για μας. Γιατί συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Ο κύριος Μάιερ χτες σε ένα άλλο πλαίσιο διευκρίνησε ότι δεν αρκεί να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα και μέσα στο χέρι μας, όχι θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε, να τα χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία. Αυτό αποτελεί ωστόσο ένα θέμα για μετέπειτα χρονική φάση. Αυτά. Ω προ το περιεχόμενο. Κάποια από τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαβουλεύσεων και στο... τα συμπεριέλαβα και στο έγγραφο εργασία. Ένα θέμα το οποίο δεν έχω αναφέρει και ίσως ε, κάποιοι να περίμεναν να το ανέφερα πρώτο-πρώτο, αλλά ε, για μένα τα θέματα περιεχομένου είναι πιο σημαντικά και πιο σημαντικά από τα διοργανωτικά ζητήματα. Είναι και, αυτό σημαντικό, ωστόσο. Θέλουμε να μείνουμε στο επίπεδο της σύστασης προς τα κράτη-μέλη ή μήπως επιθυμούμε κάποιο άλλο μέσο. Αν σωστά θυμάμαι την τελευταία συζήτηση εδώ στην Επιτροπή, η συντηρητική πλειοψηφία δεν ήταν ομοφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία των σκιωδών εισηγητών συμφωνούν μαζί μου για να καταστεί οδηγία αυτή η σύσταση. Δεν ε, θέλουμε να παραμείνουμε στο επίπεδο της σύστασης, το προαιρετικό επίπεδο, αν θέλετε. Ξέρετε τι γίνεται με τις συστάσεις. Ε, αν δεν εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη σωστά τις οδηγίες, γιατί να ακολουθήσουν τις συστάσεις. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να καταστεί νομοθετική πράξη, γιατί πρόκειται για μια καθολική υπηρεσία, θεωρώ. Και αυτή καλούμαστε να εγγυηθούμε. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός λοιπόν ο χαρακτήρας για τα να λάβει τη μορφή οδηγίας. Και αυτό λοιπόν θα μας απασχολήσει ως θέμα. Απογοητεύτηκα ιδιαίτερα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 είχε ανακοινώσει ότι προτίθετο να καταθέσει πρόταση νομοθετικής πράξης. Θεωρώ ότι η σύσταση δεν αποτελεί νομοθετικό μέσο είναι πάρα πολύ ήπιο μέσο. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και αν σωστά κατάλαβα χτες τον κύριο Μπαρνιέ, θεωρεί και αυτός ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Ενδεχομένως ε, να μην επικράτησε η άποψη αυτή μεταξύ των επιτρόπων, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει αυτή την οδό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε γιατί και αυτό ασφαλώς θα επηρεάσει και όλα τα περιεχόμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η σύσταση είναι κάτι διαφορετικό από την οδηγία και θα πρέπει με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά. Τι προτείνω λοιπόν για το μέλλον. Φυσικά θα προσπαθήσουμε με τον Μάλκομ να λάβουμε την έκθεση και συμφωνώ, αν συμφωνούν και οι σκιώδεις, να προτείνουμε ενισχυμένη συνεργασία υπό το άρθρο 50 στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία στη σύσταση τα οποία έχουν αρμοδιότητα. Μπορούμε να κάνουμε την ε, πρόταση αυτή στην ΕΚΟΝ, αλλά πάντα ε, υπό την ε, ηγεσία, θέλετε, της Επιτροπής της δικής μας, της Επιτροπής ΙΜΚΟ, να προτείνω επίσης να κάνουμε και μια ακρόαση για το θέμα αυτό, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά και οι επιστήμονες να κληθούν να παρουσιάσουν την άποψή τους, να λεφτεί και αυτή η υπόψη. Οι συντονιστές έχουν συμφωνήσει επί της αρχής για τη διοργάνωση μια ακρόαση ε, και στην παρούσα φάση προετοιμάζω ένα σχέδιο για την ακρόαση αυτή. Θα, το μεταβιβάσω στους ε, σκιώδεις για να το ελέγξουν γιατί θέλουν να υπάρξει συνεργασία να μην προκύψουν ε, τεχνητές διαφορές επειδή κάτι δεν έχει ληφθεί υπόψη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να εργαστώ. Να προτείνω βάση της ακρόασης να προβώ στην κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης εγκαίρως και αν είμαστε η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να μου δώσετε και τις δικές σας απόψεις για το κατά πόσον θα πρέπει να ζητήσουμε οδηγία ή θα μείνουμε στο επίπεδο των συστάσεων. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε εδώ και τώρα αυτό, εκ των προτέρων, αλλά θα ήθελα να, να παρακαλέσω τους κοιόδους εισηγητής να τα συζητήσουν αυτά στο συντορικό των ομάδων τους. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό, για να είναι και συνεπές το έργο μας. Και βάσει όλων αυτών να διαμορφώσουμε το τελικό κείμενο. Αυτό λοιπόν το απευθύνω ω έκκληση στους εισηγητές. Και Στη συνέχεια, σκοπός μας είναι να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Ιούνιο, προκειμένου να έχουμε αρκετό χρόνο, προκειμένου όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι εκτενέστατα, να τα συζητήσουμε εντελεχώς, να βρούμε συμβιβασμούς όπου αυτό θα είναι απαραίτητο και αυτό θα ταιριάξει πάρα πολύ καλά γιατί εξέτασα και το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής το οποίο μας και χτες γιατί ο Επίτροπος Μπαρνιέ έχει προγραμματίσει τον Ιούλιο να κάνει περαιτέρω βήματα στο θέμα αυτό. Και άρα μπορεί να το πράξει αυτό βάσει και όσων έχει αποφασίσει τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι θα δώσουμε μια σαφή υπόδειξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσει το έργο αυτό. Και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει την νομοθετική αυτή έκθεση πρωτοβουλίας την οποία θα πρέπει να εγκρίνει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Αυτά λοιπόν, αυτές οι αδρές γραμμές, πρώτες σκέψεις για τη διαδικασία τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα πρώτα να καλωσορίσω μια ομάδα κυριών από το Κάσλερ. Καλωσορίσατε, είσαστε εκεί πίσω από, τη, ε, από το κόμμα της κυρίας κάσλε. Είναι μεγάλη η αίθουσα, είστε πολύ μακριά, αλλά παρόλα αυτά σας βλέπουμε. Να πω μία πρόταση να τις καλωσορίσω και εγώ. Και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ πέρα αυτές οι γυναίκες. Uh, um, Μάλιστα. Ας ακούσουμε τώρα τις παρατηρήσεις για αυτές τις πληρέστατες προτάσεις που μας παρουσιάζει. Ο κύριος Μάιερ θα πάει πρώτο στο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Εύελιν έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα αυτό και το υποστηρίζει αυτό τα και δικαίως. Υπάρχει και αυτή η μελέτη για τον βασικό λογαριασμό, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Ήταν πολύ δύσκολη στην εκτέλεσή της. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί ακόμα μαζί της, γιατί δεν είχα το χρόνο. Αλλά βρισκόμαστε καταρχάς στο θέμα της αρμοδιότητας ε, των ε, επιτροπών και θα πρέπει να πω ότι ασπάζομαι πλήρως την άποψή σου, γιατί το θέμα δεν είναι πρόβλημα των τραπεζών, στην οποία περίπτωση ήταν αρμόδια η Επιτροπή ΕΚΟΝ, οι τράπεζες δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα γιατί δεν ε, κάνουν τίποτε που δεν επιθυμούν. Θα πρέπει να τις αναγκάσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Άρα μπορούμε λοιπόν θεωρώ να δικαιολογήσουμε την ε, αρμοδιότητά μας με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Ελευθερία για α, παροχή υπηρεσιών και ε, εμπορευμάτων και τα οποία δεν μπορώ να πληρώσω αν δεν έχω λογαριασμό ε, ελευθερία ε, έφερσης εργασία κάπου αλλού γιατί οι πιο πολλοί εργοδότες δεν θα έδιναν δουλειά σε κάποιον χωρίς λογαριασμό ελευθερία του κεφαλαίου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ροής του κεφαλαίου διασυνοριακά χωρίς λογαριασμό δεν γίνεται αυτό άρα πρόκειται για την εφαρμογή των τεσσάρων αρχών της ενιαίας αγοράς. Άρα θεωρώ ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Επίσης συμφωνώ ότι η σύσταση στο σημείο αυτό δεν πρόκειται να έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα, γιατί στη σύσταση η έννοια, ο ορισμός που χρειαζόμαστε για τον βασικό λογαριασμό δεν θα μας καλύψει η οδηγία θα είναι πιο δέουσα. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η βασική μας σκέψη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ρυθμίζουμε μόνο αυτά που είναι απαραίτητα. Όλοι τα υπόλοιπα επαφίεται στο επίπεδο της επικουρικότητας, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Αυτό ισχύει και εδώ. Χρειάζεται σαφής αλλά και απλός ορισμός για το τι μπορεί να αξιώσει ο καταναλωτής προκειμένου να υπάρχει πραγματική ενιαία αγορά. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Και οι συνέπειες ε, για τις τράπεζες αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΚΟΝ. Μπορεί να αποτελέσει συνεργασία στα συνήθη πλαίσια, η ενισχυμένη συνεργασία, αλλά ο τραπεζικό τομέα δεν αποτελεί το βασικό θέμα. Το βασικό θέμα είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Συμφωνούμε λοιπόν ω προ αυτά. Ευελίν, θεωρώ ότι αν ε, πολεμήσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια στην ομάδα, στις ομάδες μας για να καταλήξουμε χωρίς καυγάτες σε συμφωνία με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αυτά ως προς το περιεχόμενο θα συζητήσουμε αργότερα. Good. Thank you very much. Uh, so... Μάλιστα, ευχαριστούμε ο κύριος Κρόιτσμαν, Ε, του κύριος Σμιτ εξ ονόματο του κ. Σμιτ κάποιε παρατηρήσει. Ένα βασικό ε, τέτοιο τραπέζικό λογαριασμό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για του ε, πολίτε που το επιθυμούν. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε κάποιου από την εσωτερική αγορά επειδή δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό, γιατί έτσι δημιουργούμε προσκόμματα για βασικέ ε, δραστηριότητε, αποκλείουμε ακόμη και την πρόσβαση στην στέγη. Χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο πέραν κάθε αμφιβολίας θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι υπέρ και μιας οδηγίας, διότι όταν δείτε τις μελέτες του Τμήματος Πολιτικών για τις Τραπεζικές Υπηρεσίες είναι ενδιαφέρον όταν βλέπετε, Φερρυπίν, πως στο Λουξεμβούργο οι φτωχοί μπορούν να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό αλλά όσοι δεν ε, μιλάνε τη γλώσσα και το ανέφερε και η κυρία Γκέπχερτ ε, έχουν πρόβλημα ή στη Γαλλία, στην Ιταλία δημιουργούνται προβλήματα για κάποιους που θέλουν ε, να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στην έκθεση. Συζητήσαμε τον Όλε Σμιτ και βλέπετε ότι στις σημειώσεις του δεν ε, αναφέρει τίποτα για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Κανονικά δεν έπρεπε ε, να υπάρχει τέτοια ανάγκη, αλλά όταν χρειαστεί θα πρέπει να το προβλέψουμε. Φυσικά δεν πρέπει να υποχρεώνεται κανείς να ανοίγει ένα λογαριασμό, είναι προφανές. Επίσης ε, οι τράπεζες δεν χρειάζεται να προφέρουν υπηρεσίες όπως πιστωτικές κάρτες και άλλες υπηρεσίες που υπερβαίνουν έναν απλό λογαριασμό για πληρωμές. οι τράπεζες ε, θα πρέπει να ε, καλωσορίζουν τους ε, νέους πελάτες, ακόμη και διασυνοριακούς πελάτες, ακόμη και τους ανεπιθύμητους. Νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει αυτό το πολιτικό μήνυμα. Δείτε στη μελέτη ότι δεν είναι το πρόβλημα των πλουσίων αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, Μάγερ, ε, ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα εσωτερικής αγοράς. Δεν είναι αποκλειστικά αμυγός μόνο πρόβλημα των τραπεζών. Ευχαριστούμε την Εύελιν και περιμένουμε τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος, η κυρία Τούριν, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένα το ζήτημα, δεν θα δυσκολευτούμε να συμφωνήσουμε γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Με ενθαρρύνουν όλα αυτά που άκουσα. Δύο από τους δέκα Ευρωπαίους δεν έχουν πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά λένε τα στοιχεία. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Μόνο έξι κράτη-μέλη βλέπουμε ότι διαθέτουν έχουν κατοχυρώσει νομοθετικά το βασικό δικαίωμα ανοίγματο ενός ε, ε, βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Άρα χρειάζεται να κινητοποιηθούμε διότι για μας είναι θέμα αποκλεισμού κάποιων από την κοινωνία. Δηλαδή σήμερα αποκλείεται κανείς από βασικές δραστηριότητες στην κοινωνία αν δεν διαθέτει βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Δεν είναι θέμα πιστοτικών καρτών, ε, το ξαναλέμε. Ε, πρόκειται για βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Είναι βασικό δικαίωμα. Είμαστε υπέρ αυτή τη προσέγγιση λοιπόν και ε, είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα αλλάξει κάτι με τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξέδωσε το καλοκαίρι, γιατί αναφέρεται εκεί ότι πρέπει να γίνει κάτι πριν το καλοκαίρι το 2012. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις με αυτήν την έκθεση, θα δούμε αν ε, γίνεται κάτι, αν αλλάζει κάτι, αν όχι. Θα χρειαστεί να ασκήσουμε και εμεί πίεση και για να απαντήσω στην κυρία Γκέπχαρτ, ναι, όσο πιο δεσμευτικό είναι τόσο το καλύτερο, γιατί προ το παρόν δεν είναι καλή η πρόταση. Η οδηγία θα ήταν μια καλή λύση, κατά τη γνώμη μα. Αυτά προς το παρόν και περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Λέει ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος Φόξ ε, ε, είναι σκιώδης, ε, δυστυχώς απουσιάζει, αλλά μου έχει δώσει τις σημειώσεις του. Θα σας τις κοινοποιήσω πρώτον. Η βασική απέτηση για να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους καταναλωτές και τους πολίτες προσυπογράφει πλήρω το στόχο. Ξέρουμε γιατί. Η κυρία Γκέπχαρτ αναφέρθηκε σε διάφορα σημαντικά σημεία. Είναι επίση σημαντική η διάκριση ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν γενικοί όροι για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ξέρουμε ποια είναι τα βασικά, οι βασικέ 20 καταγγελίε των πολιτών ότι κάποιοι μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια ε, χώρα και είναι φερέγγενο, σε άλλες ε, δεν μπορούν. Λόγω ε, ζητημάτων ε, όπως ε, η απόδειξη της διαμονής, του τόπου διαμονής. Το ανέφερε η κυρία Κέπχαρτ. Θα πρέπει να το ρυθμίσουμε κάποιο τρόπο. Επίσης να φροντίσουμε ώστε θα πάρουμε τις εκθέσεις, τη, τα στοιχεία συγγνώμη, για τις 20 βασικές καταγγελίες των πολιτικών της έκθεσης κυρίας Μπάστος και θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση κυρίας Εγκέφχαρ, το είπε και η ίδια, πρέπει να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα, να συνδυαστούν οι δύο εκθέσεις. Τώρα, ε, όταν εξετάζει κανείς διεξοδικότερα αυτή τη ε, μελέτη του τμήματος ε, πολιτικών, βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη και άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα δεν θα συμπληρώσει ε, απαραίτητα την κατάσταση. Μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα σε κάποια κράτη-μέλη. Ο κύριος Φόξ, επίσης, επειδή έχει κάνει την έρευνα ενώ εγώ όχι, μου υποδεικνύει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, αλλά έχουμε 16 διαφορετικά είδη βασικών τραπεζικών λογαριασμών στην αγορά, Άρα όταν είδαμε την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παρότι δεν αναφέρθηκε σε μονομένες περιπτώσεις η Επιτροπή, αναρωτιέμαι μήπως αυτό το στάδιο ε, είναι πρόσφορο να κινηθούμε νομοθετικά. Μήπω θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με ένα κώδικα διοντολογία για τι τράπεζε για ε, εθελοντικού χαρακτήρα μέτρα, αντί να περιμένουμε να εγκριθεί και να υιοθετηθεί η οδηγία. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία αυτή τη πρόταση αν επιθυμούμε μια ταχεία αντίδραση σε σχέση με τα προβλήματα που παρατηρούνται. μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα μέτρα σε όλε τι τράπεζε. Αν δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενδεχομένω θα μπορούσαμε μεταγενέστερα να κάνουμε αυτό το νομοθετικό βήμα. Ε, νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα του πολίτε σε ένα πρώτο στάδιο. Λοιπόν, από πλευρά μα ε, θα δείξουμε ανοιχτό πνεύμα, θα ε, δούμε κατά πόσο χρειάζεται νομοθετική δράση, θα δούμε ε, ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα, ποιο αντίκτυπο θα έχουν και θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε κάνει μια νομοθετική προπαρασκευαστική εργασία για να έχουμε έτοιμη τη δεύτερη λύση. Ας ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη, κύριος Φιλιππέλη, ο φίλος μας έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας καλωσόρισα, θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια. Αυτά από πλευρά τη ομάδα μου. Η κυρία Ροσφάρ, Βανιό. Ντιγιόν, θέλετε κι εσείς το λόγο. Βεβαίως, είστε σκιώδης. Οπότε κατά προτεραιότητα θα σας ακούσουμε και μετά θα συνεχίσουμε το γύρο των πολιτικών ομάδων και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπου ομιλητές. Ε, θέλει κανείς άλλος να εγγραφεί στον κατάλογο. Όχι, κύριε Ντιγιόν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήμουν μέλος της ε, ΙΜΚΟ ούτε καν του Κοινοβουλίου όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή αλλά πραγματικά ε, σας συγχαίρω για τις προσπάθειες που κάνατε για να κατοχυρώσετε την αρμοδιότητα της Επιτροπής στο θέμα αυτό. Υπάρχει μια γενικότερη τάση όταν πρόκειται για τράπεζες ε, Ξαφνικά η Επιτροπή ΕΚΟΝ δηλώνει, αυτό ανακηρύσσεται αρμόδια για τι αεροπορικέ μεταφορέ είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Μετά έρχεται η Επιτροπή περιβάλλοντο για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ο, κατανα... ο ίδιος καταναλωτής είναι πάντοτε. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η Επιτροπή ΕΜΚΟ, υποθέτω ότι επιθυμούσε μια πλήρη ενοποιημένη προσέγγιση για τον καταναλωτή, το Κοινοβούλιο και άρα... Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα υψής της για την Επιτροπή μας αυτό τις αρμοδιότητες δηλαδή και επικροτούμε τις προσπάθειες που κάνετε Πρόεδρε για να ε, το ε, κοινοποιήσετε θέση μας ε, στις υπόλοιπες επιτροπές. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, είναι ισοσκελισμένη η πρότασή της. Σαφέστατα εντοπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που επιθυμούν να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Επίση, διευκρινεί γιατί έχουν έρθει διάφοροι στο γραφείο μου και μου εξηγούν ότι δεν θέλουν τραπεζικό λογαριασμό. Θέλουν μετρητά. Θέλουν να τα πληρώνουν όλα μετρητά. Ε, και νομίζω ότι πρόκειται για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και φαίνεται αυτό στο έγγραφο εργασίας ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Ε, στη μελέτη επίσης διευκρινίζεται ότι αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επί τη βάση των στοιχείων που βλέπουμε στη μελέτη και σε σχέση με τις συστάσεις, πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε νομοθετική πρωτοβουλία εν ώψη και της ανακοίνωση που θα έρθει το 2012 για να αποφύγουμε ακριβώς αυτήν την αποξένωση και να κατοχυρώσουμε την κινητικότητα των φοιτητών, παραδείγματο χάρη, που είναι ένα βασικό τους δικαίωμα, όπως είπε και η συγγήτρια. Ελπίζουμε λοιπόν να συμβάλλουμε και εμείς ε, στη δουλειά της ε, εισηγήτριας στο μέλλον. Πρόεδρος, μάλιστα, θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές. Ε, η κυρία Σανομόζε. Øh, Ευχαριστώ. Καταρχήν την κυρία Γκέπχαρτ για αυτή την έκθεση και τις προτάσεις της. Εγώ έχω δύο σχόλια να κάνω. Το πρώτο είναι ότι αντίθετα με άλλα θέματα, εδώ έχει νόημα να νομοθετήσουμε. Μια οδηγία θα ήταν ευπρόσδεκτη, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε κάποιους ελάχιστους κανόνες και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν με τη σειρά τους να προσθέσουν, αν το επιθυμούν, επιπλέον κανόνες. Πιστεύω λοιπόν πως έτσι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να έχουν πραγματική πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι πιστεύω πως είναι απαραίτητο να μπούμε σε μια συζήτηση επί της ουσίας τι θα πει να έχει κανείς πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Πρώτον, ε, μπορούμε να μιλήσουμε για το κόστος, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν όλα ένα και περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον στη Δανία, όχι άνθρωποι, ε, τράπεζες με συγχωρείτε, στη Δανία, που δεν χρησιμοποιούν ε, τον ε, λογαριασμό τους παρά μόνο μέσω κάρτας ε, και πολλές φορές κοστίζει το να κάνει κανείς ανάλυση με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε ε, για το τι σημαίνει ένας τραπεζικός λογαριασμός και ποια είναι τα δικαιώματα των τραπεζών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπούμε στο ουσία της συζήτησης αυτής, δηλαδή τι σημαίνει και πώς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους τους πολίτες σε αυτό το σύστημα. Thank you. Uh, Mr. Merci, Monsieur le Président. Ο κύριος Ροσφόρ. Εγώ συνεχίζω να λέω κάτι τα εξή σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο για, σε όσους είναι εκτός. Και λέω ότι συχνά η Επιτροπή ΕΚΟΝ κάνει μακροοικονομία, ενώ η ΙΜΚΟ κάνει μικροοικονομία. Για ορισμένου ίσω να θυμίζει τα μαθήματα, εμένα μου θυμίζει αυτά που μαθαίνω στου φοιτητέ μου, που διδάσκω στου φοιτητέ. Εμεί πρέπει να κάνουμε μικροοικονομία, δηλαδή να πούμε τι κάνει ο κάθε άνθρωπο και τι δικαιώματα έχει. Νομίζω πω αυτό είναι ένα στοιχείο που μα οδηγεί στην Επιτροπή αυτή. Δεν θέλω να επιμείνω για το γεγονό ότι πιστεύω και εγώ πω η οδηγία είναι απαραίτητη. Πιστεύω επίσης πως είναι η επιθυμία του Επιτρόπου, αλλά πρέπει να τον στήριξουν και οι υπόλοιποι Επίτροποι. Γι' αυτό. Έπειτα, από τις και ίσως και σε σχέση με τα όσα είπε η Εύλην, και ένα σημείο το οποίο νομίζω δεν υπάρχει στο κείμενο της Εύλην, ούτε στο κείμενο της Κομισιόν, δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα της πρόσβασης στη στέγαση, είναι και το θέμα της πρόσβασης στην απασχόληση. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνευ ε, σταθερής ε, διεύθυνσης. Και αυτό για να αρχίσουν να φτιάξουν, να κάνουν μάλλον έναν ε, τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να έχουν κάποια διεύθυνση. Για να τους προσλάβει κάποια κάποιο γραφείο ευρέσεω εργασία και να βρουν έστω και μια προσωρινή θέση, αν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό δεν τους προσλαμβάνουν. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια δυνατότητα ε, για να δηλώνουν τη διεύθυνση σε κάποιο τρίτο χώρο, ίσως να είναι τα δημαρχία. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ή να μπορούν να δίνουν σαν διεύθυνση τη διεύθυνση κάποιου τρίτου. το πρόβλημα που έχουμε τις τράπεζες δεν είναι ανεξάρτητο από την οικονομική κρίση. Οι τράπεζες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου καταργούν θέσει απασχόληση, έχουν πρόβλημα απόδοση και βλέπουμε πω πολύ βραχυπρόθεσμα μπορεί να το θεωρήσουν αυτό ω ένα στοιχείο δέσμευση που ασκείται, μάλλον πίεση που ασκείται πάνω του ε, συγκυριακό και όχι ως κάτι το διορθωτικό. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν έντονα από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αυτό. Και σε σχέση με το όσο είπε η Εύελιν, οι εναλλακτικέ για την επίλυση διαφορών, ναι, συμφωνώ, είναι ένα πρόβλημα του να μπορεί κανείς να έχει έναν συνομιλητή. Όταν δηλαδή ένας πολίτης μεμονωμένα δεν βρίσκει σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθεί. Και ένα τελευταίο στοιχείο ε, ο, ναι, προφανώς το θέμα της κατοικίας για ένα, άνθρωπο που δεν είναι στη χώρα του αλλά μεταβαίνει σε μια άλλη χώρα, ένα φοιτητή, έναν νέο εργαζόμενο ή κάποιον τέτοιον. Πώς να βγει λοιπόν αυτός από την παγίδα ε, δεν θα πρέπει να προβλεφθεί στο κείμενο και να πούμε πως το δικαίωμα για άνοιγμα λογαριασμού πρέπει να το έχει κάθε άνθρωπος που είναι στην στο κράτος ή, βάση περιπτώσει, που να έχει στοιχεία στη διάθεσή του που αποδεικνύει ότι είναι σοβαρός, ότι δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και λέει «Ορίστε, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, έχω να σπουδάσω ή έχω την τάδε δουλειά», να μπορεί έτσι να αποκτήσει δικαίωμα για τραπεζικό λογαριασμό. Να έχω μια κατοικία θέλω και να έχω και για να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Και είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό νομίζω. Εμείς έχουμε θίξει κάποιες πτυχές κοινωνικές, αλλά θέλω να κλείσω από την οικονομική πλευρά για την ε, δυνάμωση της εσωτερικής αγοράς πιστεύω πως δεν είναι καθόλου δευτερεύον το ζήτημα. Είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα για αυτό το δέκατο για αυτά τα εκατοστά ανάπτυξης που θέλουμε να επιτύχουμε. Η κυρία Βερνιό. Θα είμαι σύντομη γιατί ήδη υπόθηκαν πολλά και ευχαριστώ την Ευελίνη για τη δουλειά της. Προσωπικά συμφωνώ και νομίζω όλοι μας συμφωνούμε, δεν χαντίθεται πλέον το ερώτημα, ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι πλέον φυσιολογικό. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Να μην στιγματίζεται ο τάδε δίνα πληθυσμό. Και όπως είπε ο κύριος Ροσφόρ και και ο κύριος Κρόισμα προηγουμένω, πιστεύω ότι στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί επιτυχημένη κινητικότητα και ανταγωνιστική. Στάζ έρασμος, εντάξει, εκεί έχει κάνει το πιστοποιητικό του έρασμος και φαίνεται ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, φυσιολογικό να μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό εκεί όπου πάει. Με μια τέτοια νομοθεσία λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε και για το δικαίωμα της ενημέρωσης για το κόστος και τη διαχείριση του λογαριασμού. Πολλές τράπεζες ε, τη σήμερα ημέρα είναι ένας λαβύρινθος για ορισμένους καταναλωτές. Ε, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Στη Γαλλία υπάρχει μια βελτίωση στην επίπεδο διαχείριση του κόστου και τη διαφάνεια. Παρόλα αυτά όμω, κατά τη διάρκεια του έτου και κανονικά δεν προβλεπόταν έτσι, ορισμένε τράπεζε επιβάλλουν κόστη που δεν ήταν προβλεπόμενα. Δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο αυτή τη οικονομική κρίση, εφάνει ότι Ορισμένα κράτη ήταν αλληλέγγυα με τις τράπεζές τους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα κατά τη γνώμη μου και οι τράπεζες επίσης να δείχνουν στους, να δίνουν, να εξηγούν τα δικαιώματα τους στους πολίτες, ώστε να είναι και αυτοί ε, υπεύθυνοι σε σχέση με τη διαχείριση του λογαριασμού τους και μόνο μια σωστή νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Μάιερ ήταν στον καταλογό μου γιατί θέλει να επανέλθει. Και μετά και ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αναφερθώ σε αυτά που είπες και εσύ, Μάλκομ. Το θέμα είναι κατά πόσον θα πρέπει κατευθείαν να ζητήσουμε οδηγία ή θα πρέπει να επικαλεστούμε την ε, εθελούσια ρύθμιση των τραπεζών. Είναι δύσκολο το θέμα. Θα πρέπει καταρχάς να δούμε αν εθελοντικά θα ήθελαν να συμμετάσχουν οι τράπεζες, αλλά δεν θα πρέπει να μιλάμε για όλες τις τράπεζες, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν υπερβολικό με την νομοθετική μας πρόταση να υποστηρίξουμε όλες τις τράπεζες, ανεξάρτητα με το είδος ε, της τράπεζας, να προσφέρουν ένα λογαριασμό. Αυτό θα ήταν υπερβολικό. Υπάρχουν μεγάλες ε, επιχειρήσεις, μεγάλες τράπεζες, ε, οι οποίες ε, κλείνουν λογαριασμού και ανοίγουν μόνο με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι θέμα των κρατών μελών να προβούν στην ε, μεμονωμένη διαμόρφωση. Αν σε, κάποιο, σε κάποια χώρα υπάρχουν εν μέρη δημόσιες τράπεζες όπου έχουν γίνει ανάλογες συμφωνίες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών, αυτό επαρκεί. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια τέτοια ταμιευτήρια. Άρα, δεν θα ήθελα να προβλεφτεί μια υποχρέωση για όλες τις τράπεζες, γιατί δεν υπάρχουν και μονοπωλιακές θέσεις, είναι υπερβολικά, ε, αν θέλετε, διαφορετική και διαφοροποιημένη το τραπεζικό περιβάλλον. Άρα να το αφήσουμε αυτό σε επίπεδο επικουρικότητας στα κράτη-μέλη. Εμείς απλά να θέσουμε κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για τους λογαριασμούς. Για τους βασικούς αυτούς λογαριασμούς. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το ποιες τράπεζες θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό θα είναι η μεταφορά κεφαλαίου, η διεξαγωγή πληρωμών, η μισθοδοσία στους λογαριασμούς αυτούς. Αυτά, τα ελάχιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Κρόιτσμαν, συμφωνώ απόλυτα με τους ε, συναδέλφους, με τον συνάδελφο, να αναφέρουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχει κανείς ε, ένα βασικό λογαριασμό. Υπάρχει στο eBay η κάρτα PayPal για τις πληρωμές, η οποία αυτόματα χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό. Δεν είναι σαν πιστοτική κάρτα που χρεώνει στο τέλος του μήνα, εάν δεν έχει κανείς ε, τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορεί να πληρώσει. Και έτσι από το eBay αποκλείονται ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού. Γι' αυτό λοιπόν, συνάδελφε Μάιερ, κάτι θα πρέπει να κάνουμε για το πρόβλημα αυτό, αλλά στα πλαίσια της επικουρικότητας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιες βασικές αρχές. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να εγκρίνει μια μεταφορά κεφαλαίου αν δεν υπάρχει φρεγγιότητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει κάποιος λογαριασμό, είτε ηλεκτρονικά και σε ό,τι αφορά την ανάληψη χρημάτων, όπου για παράδειγμα κάποιες κοινωνικές ομάδες αδύναμες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη οι τράπεζε δείχνουν τέτοιε ευαισθησίε. θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε κάποια στοιχεία. Thank you. Uh, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Βάιλερ. σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αλλά το κατά πόσο οι τράπεζε είναι όντω τόσο ευαίσθητε για να καταλάβουν τι απαιτήσει και τι ανάγκε τη ενιαία αγορά, τι να σα πω εγώ, αμφιβάλλον. Κοιτώντα ε, την ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπω ότι 12 κρατημέλη έχουν σχετική ρύθμιση, νομοθετική ή μέσω κώδικα δεοντολογίας και 15 χώρες που είναι εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπουν τίποτε. Δεν είμαι βέβαιη λοιπόν κατά πόσον τα κράτη-μέλη και οι εκπρόσωποι του τραπεζικού κλάδου έχουν διακρίνει τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Το γεγονό ότι εμείς αναγκαζόμαστε να σπρώξουμε μια κατάσταση προκειμένου να προωθηθεί η κατάσταση στα 15 αυτά κράτη-μέλη δεν είναι απαραίτητα σημάδι ευφυΐας και οξυδέρκειας. Να παρακαλέσω τον συνάδελφο Κρόιτσμαν και εσείς και εσάς να μην πούμε σήμερα τι χρειαζόμαστε, να περιμένουμε και τη διεξαγωγή της ακρόασης, να ακούσουμε τους ειδικού. Να ακούσουμε γιατί δεν έχει συμβεί τίποτα τα τελευταία τρία χρόνια. Να συζητήσουμε με το Συμβούλιο ποια είναι η τοποθέτησή του. Δεν φαντάζομαι τα 15 κρατη που δεν έχουν οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση να μην αντιλαμβάνονται ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρξει μια οδηγία πλαίσιο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ υποχρεωτικό χαρακτήρας και να μην παραμείνει στα πλαίσια μιας αθλητικής δράσης. Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετέ οι απόψει που ακούσαμε. Να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την κυρία Κέπχαρτ. Να πω και κάτι τελευταίο. Το είπα και την περασμένη φορά. Δεν ξεχνάμε και τι τεχνολογικέ εξελίξει ε, γιατί όλοι κινούνται ε, προς έναν ε, τραπεζικό λογαριασμό ηλεκτρονικών πληρωμών και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αυτό είναι ενδιαφέρον. Η πρώτη πρόσβαση σε κάποια μορφή λογαριασμού πληρωμών περνάει μέσα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας διότι φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό τηλέφωνο και το τσίπ για πίστοση ενός λογαριασμού. Ε, πρέπει να κατοχυρώσουμε λοιπόν γενικότερα την πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες. Ε, ε, όταν Όλοι έχουν ε, πρόσβαση σε ένα βασικό ε, ε, τηλέφωνο στο σπίτι τους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και πρόσβαση σε, μια, σε ένα βασικό λογαριασμό τηλεπικοινωνιών. Και αναφέρομαι στην κινητή τηλεφωνία και κυρίως για τους νέους, διότι για αυτούς αυτή είναι η πρώτη πρόσβαση στη διαχείριση των χρημάτων τους όχι απαραίτητα ένα τραπεζικό λογαριασμό. Α μην είμαστε πολύ περιοριστικοί, υπερβολικά περιοριστικοί, γιατί ξέρετε είναι ραγδέ οι εξελίξει στον τομέα της ε, τεχνολογίας. Ε, μην ξεχνάτε και αυτά που κάνουμε για τις καθολικές υπηρεσίες. Ε, κύριε Γοσφόχ, αυτή η Επιτροπή έχει συγκεκριμένη εντολή να αναλύσει όλα τα ζητήματα που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και είναι προφανές ότι πρόκειται για βασικό δικαίωμα, όπως ακριβώς και γενικότερα η πρόσβαση στις καθολικές υπηρεσίες, η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό διευκολύνει τη γενικότερη πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες. Δεν μιλάμε για δημόσιες, για ιδιωτικές υπηρεσίες. Κύριε Παλέ, σας ε, προσκαλέσαμε στο παρελθόν για να μας παρουσιάσετε την αξιολόγηση αντικτύπου. Τώρα θα μας ενδιέφερε να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας συμβάλλουμε σε κάτι ή να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις ε, της ενδοϊπηρεσιακής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε άλλη πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μάλλον γενικόλογες παρατηρήσεις σε αυτό το στάδιο. Πρώτον, ε, Χαίρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Κοινοβούλιο για αυτό το τόσο βασικό και κέρια σημασία ζήτημα για πολλούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την ε, καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η μελέτη που έκανε το, το τμήμα ερευνών ε, του Κοινοβουλίου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ διότι λείπουν συχνά ε, οι αντικειμενικές πληροφορίες, είναι κατακαιρματισμένες, οπότε φυσικά είναι καλοδεχούμενη η μελέτη. Σε σχέση με τις ημερομηνίε που μας προτείνει η κυρία Γκέμπχαρτ και εσείς ε, για τον Ιούνιο του 2012, πιστεύουμε ότι ε, μπορούμε και εμείς να συμφωνήσουμε, περιμένουμε τις απόψεις των κρατών μελών σε σχέση με την αντίδρασή τους ως προς τη συστάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου Ιουνίου για την πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών. Ευχαριστούμε λοιπόν που συνεχίζετε τη συζήτηση κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε ε, για τις ενδεχόμενες μελλοντικέ σας προτάσεις ε, που θα έρθουν να συμπληρώσουν την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θα μπορούσαμε εξάλλου να χρησιμοποιήσουμε τις δικές σας προτάσεις αν δεν αποδειχθεί η ωφέλεια των δικών μας. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέπχαρ, του κοιόδης και όλες τις απόψεις που ακούσαμε σήμερα και ε, είμαστε φυσικά πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας στο μέτρο του δυνατού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πελέ που ήρθατε και πάλι. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τις εργασίες μας ε, και ε, όσο προχωράνε και οι μελέτες και έχουμε περισσότερα στοιχεία θα παρακολουθείτε και εσείς εξελίξεις. Σας ακούσουμε την κυρία Γκέπχαρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επαναλάβω ότι το σημαντικό είναι να φροντίσουμε οι πολίτες να έχουν δικαίωμα για έναν βασικό λογαριασμό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι να υποχρεωθούν οι τράπεζες να το πράξουν αυτό και το είπα αυτό και στην εισαγωγή μου. Το θέμα λοιπόν είναι να φροντίσουμε κάθε πολίτη που το επιθυμεί γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν λογαριασμούς δικαίωμά του, Απόφαση δική του. Αλλά όποιο το επιθυμεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ένα βασικό λογαριασμό. Και αναφέρθηκαν πολλοί λόγοι και διάφοροι συνάδελφοι, Ρομπέρ, σε κάθε περίπτωση θα συζητήσω την πρότασή σου με τις υπηρεσίες απασχόλησης. Αναφέρθηκαν λοιπόν καλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δοθεί αυτό το δικαίωμα στους πολίτες. Νομίζω ότι είπα και εξ αρχής ότι δεν θεωρώ ότι κάθε τράπεζα θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει τέτοια τέτοιου λογαριασμού. Ότι τα κράτη-μέλη, νομίζω είπα, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν πώ θα οργανώσουν αυτή την πρόσβαση. Αυτό που θέλουν να είναι υποχρεωτικό είναι να το πράξουν αυτά τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να το πράξουν αν απλά προβούμε σε σύσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε από την εμπειρία μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τυφλούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και οδηγίες, υποχρεωτική νομοθεσία που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Τι φαντάζεστε ότι θα γίνει με μια απλή σύσταση. Όπως είπε και η κυρία Βάιλερ, εξακολουθούν να υπάρχουν 15 κράτη-μέλη χωρίς νομοθεσία στον κλάδο αυτό. Και η Γερμανία συγκαταλέγεται σε αυτές. Κοιτώντα λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία, πόσα άτομα έχουν δυσκολίες για το άνοιγμα ενό λογαριασμού, σε μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15%. Μα 15% είναι πολύ πιο υψηλό αυτό το ποσοστό από ό,τι θεωρούσα. Κοιτώντα τη Γερμανία, τι γίνεται, 7% του πληθυσμού άνω των 18 ετών. Αυτό δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Δεν υπάρχει επιλογή. Στην Ρουμανία είναι 39% και 26% στην Κύπρο. Εδώ θα πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε οι, πολιτικοί, οι πολίτες στα κράτη-μέλη αυτά να έχουν πρόσβαση. Την καλύτερη επίδοση έχουν οι κάτω χώρες με 3%. Αλλά είναι γνωστέ οι κατοχώρε ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά και ότι είναι πολύ φιλικοί προ τον πολίτη σε αυτά τα θέματα και αυτό είναι, γίνεται εκ νέου σαφέ. Μία σειρά σημείων τα οποία θα συζητήσουμε ασφαλώς και θεωρώ ότι προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε κάποια σημεία. Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε. Να επαναλάβω όμως αυτό που είπε η Μπάρμπαρα ή η Κρίστελ. Να μην ε, ξεκινήσουμε κοιτώντα τι δεν θέλουμε, να κοιτάμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Να κοιτάξουμε μετά με ποια μέσα μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά που επιθυμούμε να πετύχουμε. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί την καλύτερη τακτική. Και με την ε, τακτική αυτή νομίζω ότι έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου. Διαπιστώνω ότι οι ομάδες που έλαβαν το λόγο ε, όλοι πλην ενός ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν μια οδηγία. Αυτή την οδό θα ακολουθήσω και εγώ. το επιχείρημα του κυρίου Φόξ Μάλκομ ότι αυτό θα σήμαινε κάποια καθυστέρηση αν δεν είχαμε σύσταση αλλά οδηγία. Θεωρώ ότι ισχύει το αντίθετο. Δεν θέλουμε σύσταση και μετά να συζητήσουμε οδηγία. Θέλουμε κατευθείαν να συζητήσουμε οδηγία, γιατί αν ξεκινήσει η συζήτηση, αν και όταν ξεκινήσει η συζήτηση για μια οδηγία, τον ίδιο χρόνο θα πάρει. Άρα, δυστυχώς, δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Θεωρώ ότι δεν στέκει από πολιτική σκοπιάς. Δεν συμφωνώ και λυπάμαι, Μάλικολ. Εδώ διαφωνούμε. Το αντίθετο ισχύει. Καλύτερα και πιο γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα προετοιμάσουμε. Αυτά που προετοιμάζουμε τώρα θα μπορούν να επισέλθουν στο κείμενο αργότερα. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους πληρωμής μέσω κινητού. Πολύ ωραία συστήματα αυτά αλλά χρειαζόμαστε έναν λογαριασμό τραπεζικό. Αυτό αποτελεί πάντα τη βάση. Πάντα. Ανεξάρτητα από το πώς πληρώνει κανείς, χρειάζεται ένα λογαριασμό. Και όλες αυτές οι καινοτομίες... Εσύ, Μάλκολ, με είσαι ε, μηχανικός και τα παρακολουθείς όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι δυνατά μόνο εφόσον έχει κανείς ένα τραπεζικό λογαριασμό. Και γιατί να αποκλείουμε 15% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες αυτές τις θαυμαστές δυνατότητες, εφόσον το επιθυμούν. Εφόσον επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν. Ο κόσμος του 21ου αιώνα θα φέρει πολλές καινοτομίε που θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους. Αυτό είναι το θέμα. Ε, ε, για να συνοψίσουμε. Το θέμα είναι η πρόσβαση για τους πολίτες. Αποτελεί δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε μια τέτοια υπηρεσία καθολική, θεωρώ. Ως τέτοια θα πρέπει να οριστεί. Ως καθολική υπηρεσία. Και τι σημαίνει καθολική υπηρεσία, ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να έχει την δυνατότητα, την δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, και αυτό είναι σημαντικό, εφόσον το επιθυμεί, να έχει πρόσβαση σε τέτοιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συμφωνώ ότι πρόκειται για μια ελάχιστη εναρμόνιση. Εγώ γενικά πάντα είμαι υπέρμαχος της ελάχιστης ε, εναρμόνισης και προφανώς η διαμόρφωση της νομοθεσίας θα πρέπει να επαφείται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, γιατί προφανώς και διαφέρει το τραπεζικό σύστημα και οι σχετικές ρυθμίσεις, αλλά και οι συνήθειες του κόσμου. Βλέποντας ε, πόσες τραπεζικές επιταγές χρησιμοποιούνται στην Γαλλία σε σχέση με τη Γερμανία που ουσιαστικά έχει εκλείψει το σύστημα αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη κατά πόσον θα υποχρεώσουν όλες τι τράπεζε ή κάποιο τμήμα των τραπεζών ή μια συγκεκριμένη τράπεζα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι στα χέρια των κρατών μελών. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβουμε στο σημείο αυτό. Και το θέμα λοιπόν είναι να φροντίσουμε να διασφαλίζεται αυτό το δικαίωμα. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ε, για λογαριασμό στην ε, χώρα που διαμένει κανείς, θεωρώ ότι κάθε πολίτη θα πρέπει να έχει δικαίωμα να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για ενιαία αγορά, θα πρέπει να ισχύει αυτό. Εγώ έχω λογαριασμό στην Γαλλία, παρά το γεγονός ότι δεν έχω επίσημη κατοικία στη Γαλλία. Γιατί να μην επιτρέπεται και στους άλλους πολίτες, επειδή είμαι ε, Ευρωβουλευτή. Δεν θα ήθελα να τα περιορίσουμε υπερβολικά αυτά. Το πρόβλημα προκύπτει επίσης επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικά ενιαία αγορά και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, στο θέμα αυτό, γιατί η ανάγκη να ανοίξει κανείς ε, τραπεζικό λογαριασμό σε μια άλλη χώρα από αυτή που διαμένει αποτελεί ένα πρόβλημα με τη σύσταση, με την οδηγία, ό,τι και αν προκύψει τελικά, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Προκύπτει και ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε στο μέλλον και ίσως θα μπορούσαμε και για αυτό το πρόβλημα να καταρτήσουμε έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά και πάλι θα τσακωθούμε με την ΕΚΟΝ. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες. Έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Και κλείνοντας, να εκφράσω και μία σκέψη, την οποία ανέφερε και ο Ρομπέρ, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της μικροοικονομίας. Οι πολίτες, τουλάχιστον στη Γερμανία, οι πολίτες με τους οποίους συνομιλώ, αναφέρουν ότι όλο και πιο πολύ τους δίδεται η εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη του χρήματος, της οικονομίας. Εμείς με τέτοιες έκθεσεις, εκθέσεις θα πρέπει να καταδείξουμε ότι θέλουμε την Ευρώπη των πολιτών και αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε εμείς την έκθεση και όχι η ΕΚΟΝ γιατί και αυτό θα αποτελέσει ένα μήνυμα για την Ευρώπη του χρήματος και αυτό δεν το θέλει ο πολίτης θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εκεί για να καλύψει τις ανάγκες του. Και έτσι θα κλείσω. Πολύ πλούσια ήταν η συζήτηση σήμερα. Και ευτυχώ είχαμε και τον χρόνο να το συζητήσουμε. Και αυτό δείχνει το βαθμό του ενδιαφέροντα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο. Έχουμε ένα σχέδιο για να το δείξουμε στην κυριολένε. Να πω απλώς στους συναδέλφους ότι η απόφαση θα ληφθεί από τις πολιτικές ομάδες και η επιρροή που μπορείτε να ασχίσετε στους αρχηγούς των ομάδων σας θα είναι βοηθητική για να ακούστε έτσι η φωνή των καταναλωτών. Σίγουρα η κυρία Κέπχαρτ θα υποστηρίξει την θέση μας και θα στείλει σχετική επιστολή στην ε, ομάδα της, ε, θα μπορούσε ίσως να σας τη δώσει και εσά να τη στείλετε στι δική σας, ε, στις δικές σας ενημέρωση. Και ο κύριο Μάγερ βεβαίω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Πέλη. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά για το θέμα αυτό και την επόμενη χρονιά και αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας λίγο νωρίτερα. Να σας θυμίσω ότι απόψε έχουμε ακρόαση για την έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν για την παραχάραξη και την επιβολή την τελωνιακή για τα πνευματικά δικαιώματα. Ελπίζω πως θα επανέλθετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εδώ πολύ άριθμοι. Και έχουμε και πολύ καλούς ομιλητές. Αύριο έχουμε μια δεύτερη ακρόαση για την πρόταση ευρωπαϊκής τυποποίησης. Στις 9 αύριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε.